Κυρίε και κύριοι εμπειρογνώμονε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτήν την ακρόαση που έχει διοργανωθεί από τις Επιτροπές ΠΑΤΣ, ΚΟΝΤ, ΑΦΕΤ και ΔΕΒ. Πρόκειται για μια ανακρόαση που ε, αφορά την αξιολόγηση των ε, κονδυλίων, των ταμείων αλλά και των καταπιστευμάτων που έχει αφιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, πολιτική για τους πρόσφυγες. Στόχος είναι να μελετήσουμε σε ποιο βαθμό και ιδιαίτερος από το 2000 15 σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανταποκριθεί στις μεταναστευτικές προκλήσεις με τη βοήθεια των μέσων που έχει διαθεσή της, σε ποιο βαθμό τα προσάρμοσε ή δημιούργησε νέα και συχνά κατεπηγόντως με κίνδυνο να προσθέσει μονάδες σε αυτό, σε αυτό που ονομάζουμε τον δημοσιονομικό γαλαξία. Πρόκειται για το τίτλο 4 του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή τα χρήματα που ε, επενδύονται ή δαπανώνται εκτός των συνόρων της Ένωσης. Στις 16 Μαΐου θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια κοινή ακρόαση Badge, Cont ε, και λίμπε για την αποτελεσματικότητα των ε, πόρων του τίτλου 3 που στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές εντός των συνόρων της Ένωσης. Παρακολουθούμε λοιπόν αυτές τις χρηματοπιστωτικές ροές εκτός της Ένωσης τη στιγμή που τα χρήματα αυτά δίνονται μέσω της ε, χρήσης τους επιτόπου μέχρι το τη στιγμή του έλεγχου ε, και ε, της Αποτελεσματικότητά του. Θα δούμε δηλαδή ποια διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε για την επόμενη πολυετή ε, δημοσιονομική περίοδο, δηλαδή από το 2021. Αυτή η ακρόαση έχει χωριστεί σε δύο ε, πάνελ. Ε, το ένα το μοντέλο χρηματοδότηση και εξέλιξή του και το άλλο είναι αφιερωμένο στα αποτελέσματα επιτόπου. Κάθε πάνελ θα συνεχιστεί με συζήτηση θα μπορείτε να μοιραστείτε την, ε, μαζί μας την δική σας ε, προοπτική στη διάρκεια αυτής της συζήτησης και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ακρόαση ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Χαβιέρ Γκάουζο Περμούη, που είναι αντιπρόεδρος τη Επιτροπής ΑΦΕΤ, να πει και εκείνο την του, να σα κάνει και εκείνο μια εισήγηση, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Στα ισπανικά θα τα πω. Θα είμαι σύντομο γιατί έχουμε πολλούς αξιόλογους εδώ ομιλητές και θέλω να έχουμε χρόνο να τους ακούσουμε όλου και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα το μεταναστευτικό, το θυμηθήκαμε, ότι εξακολουθεί να είναι μια τραγωδία και δεν έχει λυθεί στην Ευρώπη. Με απελπισία βλέπουμε πως ένας σκάφος με 629 άντρες, γυναίκες και παιδιά και 123 ε, ε, ανήλικες μη συνοδευόμενους από κανέναν έμεινε στα νυχτά στη θάλασσα επειδή οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκαν να δεχθούν το σκάφος στα δικά τους χωρικά υδατά. Η μεταρρύθμιση του κανονισμού για το άσυλο επίσης έχει μείνει σε νεκρό σημείο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει πρόοδο στην επόμενη διάσκεψη. Την προηγούμενη εβδομάδα όμω διαπιστώσαμε ότι υπήρξε και πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σχέδιο κανονισμού όσον αφορά τη νέα γενιά ε, μέσων εξωτερική χρηματοδότηση. Κάτι πολύ σημαντικό και στη σημερινή μα ακρόαση, να δούμε τι γίνεται με τις εξωτερικές αυτές ροές όσον αφορά τη μετανάστευση. Θέλουμε να γνωρίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα από τη διαχείριση των κονδυλίων όσον αφορά τις εξωτερικές μας σχέσεις, τι γίνεται στη μετανάστευση και πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ε, δημοκρατική εποπτεία όλων αυτών των θεμάτων. Θέλουμε επίσης ε, να ακούσουμε τα μαθήματα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, πώς αντικατοπτρίζονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συγχώνευση 12 μέσων σε ένα μόνο μέσον με συνολική κάλυψη. Πώς ε, έχει προχωρήσει αυτό. Συζητάμε εδώ και πολύ καιρό για το σχεδιασμό μελλοντικών ε, χρηματοδοτικών μέσων. Δεν ξέρουμε όμως ποια δομή θα έχουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε μεταρρυθμίσεις και θέλουμε νέα μέσα τα οποία να βοηθήσουν εξωτερική μας δράση να είναι περισσότερο συνεπής με στρατοχικούς στόχους, ευέλικτη και αποτελεσματική. Θέλουμε να διασφαλίσουμε επίσης ότι η απλοποίηση δεν θα γίνει σε βάρος της διαφάνειας ή της λογοδοσίας. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε εσείς να μας πείτε λοιπόν για όλα αυτά. Πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Ελιζαμπέτ Κολέτ που είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Ευρώπη για τη Μεταναστευτική Πολιτική μετά τον Κρίστιαν Λέφλερ που είναι αναπληρωτής ε, Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, μετά τον κύριο Κούν Ντούν, ο οποίο είναι από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, και τέλο τον κύριο Ποπόφσκι, ο οποίο είναι αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη Πολιτική Γυτνίαση, τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ δηλαδή. Όπω ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι περιορισμένος ο χρόνος ομιλίας. Γι' αυτό ε, θέλουμε να ζητήσουμε από τους ομιλητές να περιορίσουν τις παρεμβάσει τους σε 7 λεπτά ο καθένας. Και χωρί άλλη καθυστέρηση δίνω το λόγο στην κυρία Κολέτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα κάνω κάποιες γενικές σκέψεις για τις εμπειρίες των τελευταίων ετών και το τι θα γίνει από εδώ και μπρο για την χρηματοδότηση της εξωτερικής διάστασης γνωρίζοντας ότι άλλοι πανελίστες έχουν μια πολύ ευρύτερη εικόνα του πώς λειτουργήσε αυτό τα τελευταία χρόνια. Η δουλειά μας βασίζεται σε κάποια έρευνα που έχει κάνει ένας συνάδελφος στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε κάποια ανάλυση του προϋπολογισμού και σε διαφορές στρογγυλές τράπεζες ε, που κάναμε για να αντιληφθούμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιείται το ΠΔΠ στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Εν ολίγης, μια περίοδο πειραματισμού και καινοτομία όσον αφορά την μετανάστευση και την ε, χρηματοδότηση και καταλητική βεβαίως λόγω της κρίσης του 2015-16 όλοι το θυμόμαστε και είδαμε σημαντική αύξηση και εσωτερικά και εξωτερικά μέσω διαφόρων ταμείων στα μέσα του 2017 ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε για να δοθούν 3,9 δις επιπλέον και 1,39 από αυτά πήγε στις αιτίες της μετανάστευσης και αυτό εν μέρη έγινε μέσω της χρήσης κονδυλίων που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αλλά και την χρήση αποθεματικών ανάγκης. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αυτά τα ζητήματα πλέον έχουν αυτά, αυτές οι πηγές χρηματοδότησης έχουν εξαντληθεί όσον αφορά την γρήγορη αντίδραση στις αλλαγές γιατί και επιπλέον ε, ευελιξία του κοινοτικού προπολογισμού έχει εξαντληθεί αλλά Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά το ότι φαίνεται ότι υπάρχει δραματική αύξηση μέσω των διαφόρων ταμείων για τη μετανάστευση, η χρηματοδότηση αυτή ε, κατ' ουσίαν πέρασε, μου είπαν, ε, πέρασαν τα κονδύλια μέσα από ένα πλυντήριο, δηλαδή έρχονταν από διάφορες πηγές να σα δώσω ένα παράδειγμα. Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έδωσε η Κομισιόν για την Τουρκία στην, το 2015 ε, ήταν από άλλα κονδύλια που ήταν ήδη ε, για την ε, Τουρκία. Οπότε κάποια από αυτά τα λεφτά τα μετράμε με διάφορους τρόπους αλλά είναι τα ίδια χρήματα και πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη όταν προσπαθούμε να αντιληφθούμε πόσα κονδύλια εξόδευονται. Πέρσι ένα ζήτημα το οποίο αντιληφθήκαμε ήταν το πως λίγοι άνθρωποι εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είχαν μια συνολική αντίληψη της λειτουργίας των ταμείων. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα γίνεται πλήρως αντιληπτό. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι ακριβώς καινοτομία ε, όσον αφορά τα νέα ταμεία όπως το Ταμείο Μαντάντα που αφορά α, ε, τους α, ε, Σύριους πρόσφυγες σε γειτονικέ χώρες και βεβαίως και το μέσο για την Τουρκία που πήγε μαζί με την δήλωση Και όλα αυτά βεβαίως έχουν βρει κονδύλια από διάφορα μέσα και συνεισφορές από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα τα ταμεία γιατί έτσι υπάρχει οικονομία κλίμακας και γρηγορότερη εκταμείευση. Παραδείγματος κάνει το μέσο για την Τουρκία έχει προγραμματίσει 2,9 δις και έδωσε έργα 1,9 δις και εκταμείευσε ήδη 900 εκατομμύρια το 16-17. Δηλαδή οποιοδήποτε γνωρίζει τα της κοινοτική χρηματοδότησης αντιλαμβάνεται ότι είναι εξαιρετικά γρήγορο. Δόθηκε έμφαση στην χρηματοδότηση, την γρήγορη χρηματοδότηση. Ε, Βεβαίω μετά το ζήτημα είναι τι συνέχεια δίνεται να υπάρχει αποτελεσματική δαπάνη όταν γίνεται γρήγορα η εκταμίευση. Όσον αφορά τώρα στον διαμοιρασμό κονδυλίων. Κάποια κράτη-μέλη καθυστέρησαν, κάναμε τις συνεντεύξεις και Ρωτήσαμε γιατί υπήρχε αυτός ο δισταγμός και υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Ένα είναι ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις έχουν δικές τους υπηρεσίες που εργάζονται επί τόπου. Ήδη ακριβώς είχαν μια τέτοια χρηματοδότηση. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι είχαν ήδη συνεισφέρει στα κοινωτικά ταμεία και δεν στα για διπλή χρηματοδότηση, αλλά όπως και με τον κοινοτικό προπολογισμό, πολλά κράτη-μέλη τώρα δεν έχουν λεφτά, προσπαθούν να βρουν κονδύλια για να ξοδέψουν και σε αυτόν τον τομέα. Και βέβαια το σημαντικότερο τώρα είναι ακριβώς να δούμε τις περαιτέρω εξωτερικές δράσεις που εστιάζουν κυρίως στις ε, γειτονικές ε, χώρες και άλλα τα κρατημέλη που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις ε, δεσμεύσεις αυτές. Άλλα ζητήματα αφορούν ε, τους περιορισμούς ε, των δαπανών καθώς 90% της εξωτερικής βοήθειας πρέπει να είναι αναπτυξιακή βοήθεια προς το εξωτερικό. Τότε έχουμε διάφορους στόχους και στον τομέα ασφαλείας που περιορίζει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει τον βασικό της στόχο. Όταν λοιπόν κοιτάμε το ποιος χρηματοδοτείται, υπάρχουν ερωτήματα για τις διάφορες υπηρεσίες και το πώς λειτουργούν, αλλά θα ήθελα να φερθώ σε κάποια σημεία ε, τα οποία αντλήσαμε από την έρευνά μας. Ε, το πρώτο είναι το σκεπτικό. Μπορούμε να σκεφτούμε για το σκεπτικό της ε, διαχείρισης της μετανάστευσης στο εξωτερικό και το πώς ορίζεται. Πρώτα απ' όλα η αιτία, οι ρίζες μετανάστευσης, η λέξη, οι, οι ρίζες μετανάστευσης πραγματικά δεν θέλω να την ξαναδώ αυτή τη φράση, δηλαδή οτιδήποτε αφορά την η βοήθεια μπορεί να πει ακριβώς ότι απευθύνεται στις αιτίες της μετανάστευσης και υποτιμά θα έλεγα και το αποτέλεσμα που έχει αυτή η χρηματοδότηση. Και τώρα γνωρίζουμε, νομίζω ότι ε, αυξημένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεν σημαίνει μειωμένη κινητικότητα από αυτές τις ε, χώρες και υπάρχει ακριβώς αυτό το λεγόμενο άλμα της ανάπτυξης, δηλαδή όσο αυξάνονται τα εισοδήματα τόσο περισσότερο φεύγει ο κόσμος. Ε, ίσως όχι προς την Ευρώπη, αλλά γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Αλλά υπάρχει και μία πιο περίπλοκη σχέση και με τους τόπους, ε, τις συνήθειες ε, της μετανάστευσης. Είναι κομμάτι των οικονομιών, και ακριβώ κομμάτι του αφηγήματο κάποιων γενεών σε κάποια μέρη, ενώ σε κάποια άλλα δεν είναι. Δηλαδή το τι κάνουμε σε μια κοινότητα, σε, μια, σε ένα μέρος του κόσμου μπορεί να μην λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Και πρέπει να μπούμε στις ε, περιπλοκότητες με αυτό το οποίο λέμε αιτίες και να προσπαθήσουμε ακριβώς να τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλούς και αντικρούμενους στόχους όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτή, ε, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας και τους ε, στόχους της ε, ανθρωπιστικής ανάπτυξης. Υπάρχει μια υποχρηματοδότηση ανθρωπιστικών κονδυλίων, ε, ε, μια αύξηση διαχείρισης ε, των συνόρων, κάτι το οποίο ο κόσμος του τους εμποδίζει να λειτουργήσουν στην τοπική οικονομία. Πώς ακριβώς λοιπόν τελικά η διαφορετική αυτή στόχη ενισχύουν ένα τον άλλον αντί να τον υπονομεύουν και ακριβώς να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προλαμβάνει αντί να αντιδρά μόνο και το νέο ταμείο που έχει συσταθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τις τελευταίες εβδομάδες ε, μας δείχνει ότι ακριβώς ε, σκεφτόμαστε και σε κονδύλια τα οποία δεν έχουν ακόμα κάπου διατεθεί ειδικά εάν μιλάμε για διαμερισμό κονδυλίων το ε, μεγάλο αυτό κουβά των 89,5 δισεκατομμυρίων ε, αναπτυξιακής βοήθειας και γειτονία, ποιος θα τα διαχειριστεί φαντάζομαι θα γίνει εκεί πέρα καυγάς ε, για το ποιος θα το κάνει αυτό αλλά το να το αντιληφθούμε αυτό και την σχετική λογοδοσία νομίζω είναι κάτι το πολύ βασικό όσον αφορά τα διδάγματα από τα κονδύλια είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία αλλά κάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το να προσπαθούμε ακριβώ ε, να δούμε το τι έχουμε μάθει και το ποια είναι τα μέτρα της επιτυχίας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε πολύ ε, χοντρικά μέσα, δηλαδή ποσοστό επιστροφών σε συγκεκριμένες χώρες και το επίπεδο ροών προς την Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε κάποια μέτρα της επιτυχίας, να αντιληφθούμε το τι σημαίνει επιτυχία, τι προσπαθούμε να πετύχουμε και πώς θα το μετρήσουμε μακροπρόθεσμα και στο πλαίσιο αυτό νομίζω πως υπάρχει μια ευκαιρία να γίνουν γρήγορα οι αξιολογήσεις για το πώς πηγαίνουν οι δαπάνες γιατί οι αξιολογήσεις θα είναι έτοιμες ε, τη δεκαετία του 2020, οπότε δεν θα προλάβουμε τον προπολογισμό. Πρέπει να το δούμε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Ξέρετε ότι οι διερμηνείς βρίσκονται σε διένεξη με την δίκηση, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το ωράριο που είναι μέχρι τις 6 και 30. Οπότε οι εμπειρογνώμονες παρακαλώ 7 λεπτά ο καθένας, όχι παραπάνω. Ο δεύτερος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Κριστιό Λεφλέρ. Παρακαλώ. Mm. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο σε αυτά που έχω να πω. Θα περιοριστώ σε μερικές μόνο παρατηρήσεις όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής μέσα στο οποίο εντάσσεται η εξωτερική διάσταση της χρηματοδότησης για την μετανάστευση. Έτσι κι η ΔΕΦΚΟ και η Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν διαπιστώσαμε νομίζω ότι υπήρχαν ε, εξελίξεις προς μια πιο συνολική αντιμετώπιση της μετανάστευσης όσον αφορά σχέσεις μας με τρίτες χώρες και άλλες περιοχές του κόσμου. Δημιουργήθηκαν νέες εταιρικέ σχέσεις, υπογραμμίστηκε επίσης η επιμερισμένη ευθύνη για το θέμα. Επίσης, και το ακούσαμε ήδη όσον αφορά τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, υπήρξε το Trust Fund, το καταπίστευμα, υπήρξε η χρηματοδότηση προς την Τουρκία, υπήρξε το πλαίσιο επίσης εταιρική σχέσης με διάφορες χώρες της Αφρικής και άλλες επίσης περιφερειακές προσεγγίσεις με άλλα μέρη του κόσμου, με το Αφγανιστάν για παράδειγμα, όπου έχουμε συμπεριλάβει και την μετανάστευση ως μία διάσταση της συνολικής μας σχέσης με αυτή τη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση αρχίζει να αποφέρει κα... καρπούς. Είναι βέβαια μια διαρθρωτική σχέση που δεν φέρνει τα αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ποια είναι η συνεργασία και μετά να περιμένουμε για αποτελέσματα. Πάντως υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τρίτες χώρες, όσον αφορά τη μετανάστευση, ε, με τρόπο που να ταιριάζει στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές και οι προσδοκίες και οι ελπίδες επίσης. Πάντως βλέπουμε ότι και οι εταίροι μας και σε διμερές επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό ευαισθητοποιούνται όλο περισσότερο και σε πολυμερές επίπεδο και το δείχνουν αυτό στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ μας. Έχουμε ένα σαφές παράδειγμα που είναι οι σχέσεις μας με την Αφρικανική Ένωση και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης όπου διμερός και μέχρι το Πιτζάν πέρυσι προετοιμάσαμε έναν αντιπυρωτικό διάλογο προσπαθώντας να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν στην Αφρική, στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ των δύο πλευρών. Και αναπτύξαμε και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ένα τριμερές πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Και γενικά, μιλώντας, αλλά και πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της Λιβύης, όπου εκεί όλοι οι παράγοντες δεσμεύτηκαν. Η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διάφορες υπηρεσίες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ. Θελήσαμε ευέλικτη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Trust Fund και υπήρξαν αποτελέσματα αυτά από τον Εύριο-Δεκέμβριο που μας πέρασε. Συνεχίζεται βέβαια η δουλειά και επεκτείνεται με τις ε, λιβικές αρχές προκειμένου να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη λαθροδιακίνηση. Σε επίπεδα τεχνικό, ε, ανώτερων αξιωματούχων. Είχαμε πολλές επαφές με τις λιβικές αρχές και θα συνεχιστεί στην πρώτη περίπτωση πριν από το καλοκαίρι, στη δεύτερη μετά το καλοκαίρι. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια για τις αιτίε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε και ο Προλαλήσας, προλαλήσας μάλλον, ότι δηλαδή το να αντιμετωπιστούν οι αιτίε. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε την απτυξιακή βοήθεια τα τελευταία 50 χρόνια, χωρίς όμως να είμαστε ιδιαίτερα επικεντρωμένοι. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την υλοποίηση του καταπιστεύματος, του κατασματικού αυτού ταμείου, ε, προσπαθούμε να έχουμε μια προσέγγιση πιο λεπτομερή, κοιτώντας τα αποτελέσματα της κάθε δράσης μας. Και συγχρόνως προσπαθούμε να έχουμε και μια πιο συνολική ανάλυση του τι ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στο μεταναστευτικό. Εδώ μια λέξη κλειδί είναι η ένταξη, αλλά αυτή η λέξη μπορεί να σημαίνει πολλά. Συνήθως είναι οικονομική, κοινωνική, αλλά εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είναι και πολιτική. Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή των κοινοτήτων τους, των χωρών τους, να νιώθουν δηλαδή ότι είναι τους δίνεται η ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον τους και το μέλλον της χώρας τους. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Τώρα συνεργαζόμαστε προκειμένου να υπάρξει μια πιο πλήρης οικονομική αντιμετώπιση στα πλαίσια του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα βέβαια το μεταναστευτικό με την κάθε χώρα εταίρο. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε δράσεις και χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό, να συμπεριλαμβάνεται δηλαδή σε κάθε είδους δράση που έχουμε με τις διάφορες χώρες του κόσμου. Και όπως φαίνεται και από τις προτάσεις που υποβάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, αυτό γίνεται περισσότερο ε, βλέποντας την μετανάστευση συνολικά Ακριβώς επειδή το μεταναστευτικό συνδέεται τόσο πολύ με ένα σωρό άλλα, άλλες μορφές σχέσεων που έχουμε με τους εταίρους μας. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντούνς. Euh, Θα προσπαθήσω να τα πω τόσο καλά όσο και ο Κριστιαν που ε, μίλησε μόνο 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφραστώ για ένα θέμα ε, που είναι πολύ σημαντικό για την αναπτυξιακή πολιτική. Ε, άρα λοιπόν η προτεραιότητα που είναι η μετανάστευση έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο που δουλεύουμε και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο νέο έγγραφο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης την Ευρωπαϊκή Συνένεση και ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ Ε, θα περιοριστώ σε κάποιε γενικέ παρατηρήσει που αφορούν τα θέματα που σα ενδιαφέρουν. Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι όταν βλέπουμε την ε, μετανάστευση με τα αναπτυξιακά μα μέσα, ανέκαθεν καθοδηγούμεθα από δύο βασικέ αρχέ. Η πρώτη είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε και επιλέγουμε από αυτό που ο πρόεδρος αποκάλεσε το δημοσιονομικό γαλαξία, φυσικά όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα πάντοτε το κάνουμε ε, με βάση την εντολή τους. Αυτό ήταν θεμελιώδου σημασία γιατί θέλουμε να εργαζόμαστε με σε πλήρη σεβασμό της νομικής βάσης με τις δυνατότητες αλλά και με τους περιορισμούς των δημοσιονομικών μας μέσων. Δεύτερον, οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται σε συνεργασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Συνεργασία χωρίς εταίρους, ε, ε, δηλαδή ε, να λαμβάνουμε υπόψη το γεωγραφικό πλαίσιο εντό του οποίου εργαζόμαστε. Αυτή είναι η δεύτερη βασική μας αρχή που έχουν μεταφραστεί αυτές οι αρχές σε δυο τρει βασικά ζητήματα. Πρώτον, αφορά τι κάνουμε ακριβώς. Αυτό ξεπερά την Αφρική, εφαρμόζεται παντού, αλλά με την Αφρική έχουμε το παράδειγμα της, της δήλωσης της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε εκεί. Ε, δηλαδή συνολική, ευρεία και ισορροπημένη προσέγγιση για την ε, μετανάστευση. Και αυτό βρίσκεται στην καρδιά των όσων κάνουμε για όλα τα θέματα της μετανάστευσης. Ε, εξετάζουμε τις, τα αίτια ε, μπορεί να είναι βαθύς όρος, αλλά είναι και πολύ σκόπιμος, γιατί όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, ε, την τακτική, την, άτακτη και την μετακίνηση, αυτό το οποίο οδηγεί τον κόσμο να φύγει από το σπίτι του και από την κοινότητά του, που δεν είναι κάτι το προτιμά κανείς, και, αλλά αναγκάζονται να μετακινηθούν ε, Χρειαζόμαστε όμως πιο λεπτομερή ανάλυση των αιτίων. Δεύτερο θέμα σχετίζεται με την νόμιμη μετανάστευση. Ε, υπάρχουν, ε, γίνεται πολύ νόμιμη μετανάστευση ε, στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και αυτά τα νόμιμα πλαίσια μετανάστευσης στην Αφρική τα έχουμε στηρίξει και στην Ασία επίσης. Σε τρίτον, υπάρχει το ζήτημα των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί μέσα σε κάποια περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που βλέπουμε στο κέρας της Αφρικής. Τα μεγαλύτερα, οι μεγαλύτεροι καταφλισμοί προσφύγων είναι στο κέρας της Αφρικής, είναι το Νταχάμπ. Βλέπουμε ότι ε, Πολύ λίγοι από αυτούς τους πρόσφυγες φτάνουν στην Ευρώπη γιατί, γιατί φιλοξενούνται ε, με όσο γίνεται πιο ανθρώπινο τρόπο στην περιοχή τους και ε, στηρίζουμε τις χώρες, ε, τις κοινότητες που υποδέχονται και τους εκτοπισμένους πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει και για το Αφγανιστάν, μέσα στη χώρα την ίδια, αλλά και στις γειτονικέ χώρες όπου στηρίζουμε την αυτονομία και την αυτάρκεια ε, των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σε μετακίνηση των προσφύγων και των ε, εσωτερικά εκτοπισμένων. Έπειτα θέλουμε να διακόψουμε και να σπάσουμε αυτό το μοντέλο ε, business που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι και οι διακινητές. Αν δούμε όμως τι κάναμε στην Αγκαντές, όπου πολλοί κόσμος ε, στην ουσία έχει κάνει δουλειά του αυτό το πράγμα. Προσφέραμε λοιπόν εναλλακτικέ, προσφέραμε, ε, δουλέψαμε στην τοπική οικονομία για να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο ευημερία για αυτόν τον κόσμο και αρχίζουμε να βλέπουμε αλλαγέ επιτόπου. Λοιπόν, ε, έτσι ε, όλα αυτά μεταφράστηκαν σε ένα επιχειρησιακό εργαλειοθήκη μάλλον που ο Χριστιαν τον έφερε ήδη και διάφορα μέσα έχουμε, το πιο σημαντικό βέβαια είναι είναι το καταπίστευμα το ευρωπαϊκό. Τέλος, για τα αποτελέσματα γιατί είναι σημαντικό αυτό για μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ερευνητική δυνατότητα που συνδέεται με συγκεκριμένες γεωγραφικές καταστάσεις και θέλουμε να καταλάβουμε μέσω της συνεργασίας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ποια είναι τα βασικά αίτια, τι λειτουργεί επίσης και τι δεν λειτουργεί. Έπειτα, φτιάξαμε ένα σύστημα παρακολούθησης και διδαχής, δηλαδή πέρα από τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που κάνουμε εμείς, έχουμε έτσι και εξωτερικές εκθέσεις. Η πρώτη μάλιστα είναι διαθέσιμη στο ε, website του Ευρωπαϊκού Καταπιστεύματος και τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης είναι θετικά για το πώς καταφέραμε μέσα από τις ενεργειές μας να ε, απευθυνθούμε στις ε, κοινότητες υποδοχής, να στηρίξουμε την τοπική διακυβέρνηση, στις διευθυντικές προσεγγίσεις και να συνδυάσουμε σύντομη δράση με μακροχρόνιες στρατηγικές. Τέλος για τα αποτελέσματα και ελπίζω πως η Λίντα Μακάβανα αργότερα θα επανέλθει σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουμε συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή Ανάπτυξης, Έγινε μια αναποστολή από την Επιτροπή αυτή στην Ουγγάντα και τη Σενεγάλη και από ό,τι κατάλαβα όντως το αποτέλεσμα αυτής της ε, αποστολής ε, που από τους ε, ευρωβουλευτές ήταν θετικό για να, γιατί κατάλαβαν καλύτερα τι κάνουν και κατάλαβαν ότι πόσο, πόσο κέρυες είναι αυτές οι δράσεις μας και ποια ακριβώς είναι τα διμερεί προγράμματα που χρηματοδοτούμε. Και και έτσι βοηθήθηκε και ο διαστατικός διάλογος με τον Επίτροπο Σουίσα. Μάλιστα. σχαρτήρια Έξι λεπτά και 59. Ο κύριος Ποπόφσκι. Ε, ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο σύντομος. Η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια αναδρομή στα τελευταία τρία χρόνια και να λύσουμε κάποια διδάγματα γιατί πράγματι το 2015 δεν αλλάξαμε μόνο την προσέγγιση μας όσον αφορά τα κονδύλια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε και αυτό ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν γιατί ακριβώς τα νέα μέσα πήγαιναν πολύ πιο πέρα από οτιδήποτε μπορούσε να κάνει ο προπολογισμό. Καταφέραμε λοιπόν να συνδέσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης με την χρηματοδότησή μας για τη μετανάστευση. Τα εργαλεία αναφέρθηκαν, το καταπίστευμα για την Αφρική, το μέσο για την Τουρκία, το καταπίστευμα για την Συρία, ειδικά η πιο κοντινή μας, στην πιο κοντινή μας γειτονιά, σε στενή συνεργασία, ειδικά και στις χώρες προέλευσης και διέλευσης και προορισμού. Εστιάσαμε στον διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου από την Βόρεια Αφρική με το καταπίστευμα για την Αφρική με βεβαίως Μέση Ανατολή μέσω του μέσου της Τουρκίας και τις γειτονικές χώρες της Συρίας, Λίβανο, Ιορδανία κτλ. Μέσω του καταπιστευματός για την Συρία. Νομίζω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε κάποια καλά αποτελέσματα δεδομένων χρονικών περιορισμών. Βεβαίω έχουμε την κατάσταση στη Λιβύη που μας απασχολεί όλους, οι ηγέτες μας το συζητούν τακτικά, εστιάζουμε στην προστασία των ε, προσήγων επιτόπου, εθελοντικές επιστροφές, ε, την κατάσταση στη Λιβύη. Ένα παράδειγμα, 22.000 εθελοντικές επιστροφές έγιναν μέχρι στιγμής. Σημαντικός αριθμός, ε, παρά το ότι ο συνολικός αριθμός των προσήγων και μεταναστών στη χώρα είναι ακόμα πολύ ψηλός. Το μέσο για την Τουρκία καταφέραμε να το εφαρμόσουμε πάρα πολύ γρήγορα 3 δισεκατομμύρια μέσα σε δύο χρόνια ξοδέψαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 17 τώρα έχουμε την επόμενη δόση τα αποτελέσματα είναι χαρακτηριστικά γιατί καταφέραμε να δώσουμε άμεση βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες από τα 3,5 εκατομμύρια που ζουν στην Τουρκία και υπάρχουν απτά ωφέλη όπως 125 ε, σχολεία, σύν άλλα 50 προκατασκευασμένα και στο μέλλον βεβαίως θα περάσουμε σε πιο κοινωνικο-οικονομική στήριξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, ένταξη των Συρίων στην αγορά εργασίας Τουρκίας, στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε Ιορδανία και Λίβανο, εστιάζουμε σε βιωτικέ συνθήκες, αλλά και εκπαίδευση και υγεία στις κοινότητες που φιλοξενούν. Δίνουμε παραδείγματα έργων, αλλά βεβαίως αυτά αφορούν ανθρώπους και πρέπει να, τα έχουμε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εστιάζουμε ειδικά στη νέα γενιά, δεν θέλουμε να υπάρξει μια χαμένη γενιά. Και πάλι ένα παράδειγμα, το, παράδειγμα, το ποσοστό των παιδιών που πάνε σχολείο. Μιλάμε για 600.000 νεαρούς, ήδη πολύ εντυπωσιακό και αυξάνεται ο αριθμός και αυτή τη στιγμή υπάρχει και κάτι άλλο. Μια εκδήλωση αυτή τη στιγμή στην Φλαζέ ε, την πλατεία εδώ των Βρυξελών όπου οι Σύριοι λένε το πώς ε, άλλαξε η ζωή τους μέσω της ε, στήριξης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. ξεκινήσαμε το 2015 μετά έπρεπε να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Επεκτάθηκε και η γεωγραφική κάλυψη, οπότε τώρα το καταπίστευμα λειτουργεί και στην Αρμενία και στα Δυτικά Βαλκάνια επεκτείνουμε ακριβώς ε, το μέσο αυτό ανέφερα τη δεύτερη δόση των 3 δισεκατομμυρίων που ελπίζουμε να ξεκινήσει αργότερα φέτος και έχουμε φτάσει σε υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης στο βορειοαφρικανικό παράθυρο το λεγόμενο ο τρέχον προπολογισμό είναι στο επίπεδο των 524 εκατομμυρίων ήρθαμε σε επαφή και με το Κοινοβούλιο και με μεγάλη μου χαρά φιλοξένησα και εσάς κύριε Πρόεδρε στην συνεδρίαση της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής και δικαίως βεβαίως και στο μέλλον αυτή η σχέση θα γίνει πιο έντονη με την έννοια ότι ο κανονικός ε, Ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων για τα μαθήματα του ΠΔΠ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο κ. Λεφλέρ. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις στο προτινόμενο νέο μέσο και έχουμε ένα στόχο δαπάνη σε 10% στη μετανάστευση συν ένα αποθεματικό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ακριβώς για να ανταποκριθούμε στην μεταναστευτική πίεση θέλουμε ακριβώς να υπάρχει μια ευελιξία και να μπορούμε να αντιδράσουμε με κάτι το οποίο δεν υπήρχε όταν αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να στηθεί μια τελείως νέα δομή για να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καταφέρατε, συγχαρητήρια. 6 και 22. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τους βουλευτές. Η κυρία Βερζιά. Ναι, ναι, συγγνώμη, αργότερα. Ε, είδα ότι είναι το όνομά μου. Μια ε, ερώτηση είναι για τον Κριστιαν Λεφ, γιατί αναφέρατε όλα τα καινούργια προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν η πρωτοβουλία για το, της DG Home μιλήσατε για την εξωτερική πολιτική. Πώς η εξωτερική πολιτική θα αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι μάλλον σχόλιο. Σε σχέση με την διάσκεψη κορυφής του Αμπιτζάν. Κοιτάξτε, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στη συμφωνία στο Μπιτζάν στα τελευταία στάδια. Δηλαδή, δεν ήμασταν καν κοντά, ούτε είπαν ότι «Α, τέλεια ιδέα και θέλουμε να συνεργαστούμε». Όχι, αντίθετα υπήρχαν πολλά προβλήματα για συμφωνία και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς στι εκτιμήσεις μας για το τι συμβαίνει επί τόπου. Διερωτώ με αν ξέρω πως δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Υπουργό από τον ε, Νίγηρα το ίδιο ειλικρινής θα πρέπει να είμαστε και για την τελευταία μου παρατήρηση. Τι έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει διάφορα. Και είδαμε στην Ουγκάντα όταν είχαμε τη δεύτερη συνεδρίαση επιτόπου, αλλά για την πολιτική γειτονία. Ξέρουμε πως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα για την εκπαίδευση σε όλη την περιοχή. Το είπαμε νομίζω. Θεσπίσαμε το ένα στόχο ώστε κάθε παιδί στην Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία στους προσφυγικούς καταβλισμούς θα πήγαινε σχολείο μέχρι το Σεπτέμβριο πέρυσι. Αλλά αυτό δεν το πετύχαμε και το ξέρουμε. Όταν κάνουμε τέτοιου είδους παρουσιάσεις λοιπόν, καλό θα ήταν να ξέρουμε στοιχεία για το πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Πρόκειται για πολύ πολύ δύσκολα πολιτικά ζητήματα. Πολύ δύσκολες πολιτικές επιλογές πρέπει να γίνουν. Ένα από τα προβλήματα εξ αρχή σε αυτή την υπόθεση της μετανάστευσης είναι ότι τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε σημείο που και ακόμα και η ΑΕΑ δεν ήξερε τι ακριβώς γινόταν. Και αυτό είναι θέμα. Μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις για το τι να κάνουμε με τα χρήματα θα έπρεπε να λαμβάνονται από τις δημοσιονομικές αρχές, δηλαδή Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, γιατί ποιο λαμβάνει τι στρατηγικέ συζητήσει να φτιάξει όλα αυτά τα ταμεία και πότε λαμβάνει αυτή η απόφαση κάθε φορά. Είναι δύσκολο. Συγκεντρώνονται, το ένα συμβούλιο ακολουθεί το άλλο, ε, αλλά δεν ενημερωνόμαστε πάντα το εδώ. Εμείς τρέχουμε από πίσω να δούμε τι γίνεται. Στο μελλοντικό σχεδιασμό λοιπόν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει περισσότερο στις στρατηγικές συζητήσεις. Και έπειτα, πιο ειλικρινή αξιολογή για την κλίμακα του προβλήματος μέσω κοινή δέσμευση, καλύτερη κατανόηση, λιγότερες παρανοήσεις όσον αφορά το, το πλαίσιο τη πολιτική τη Ένωση στο μέλλον. Κυρία Βερυζιά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω λίγο ε, ε, μια ανακοίνωση. Στις 19 Ιουνίου σήμερα, αύριο είναι η μέρα των προσφύγων. Οι διάφορες οργανώσεις δίνουν τα στοιχεία που έχουν για τους πρόσφυγες. Σήμερα πήραμε λοιπόν το ε, έγγραφο της ΥΠΑ της του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τι λέει, ε, χαιρόμαστε που για δεύτερη συνεχή χρονιά η μεταναστευτική πίεση μειώνεται. Ο αριθμός της διεθνούς προστασίας έχει, έχει κατέβει κατά 44% στην Ένωση και το ποσοστό αναγνώρισης κατά 14% έχει φτάσει στο 50%. Εν τω μεταξύ όμως τι γίνεται με την παγκόσμια κρίση η παγκόσμια κρίση των προσφύγων αυτή συνεχίζει και επιθυνώνεται. 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί πέρυσι. Ένας άνθρωπος κάθε δύο δευτερόλεπτα. Και αυτό που αυξάνεται είναι πλέον ο αριθμός των προσφύγων και όχι ο αριθμός των εκτοπισμένων, των εσωτερικά εκτοπισμένων συν 2,9 εκατομμύρια από το 2016 μέχρι το 2017. Το 85% αυτών γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, 90% ανάμεσα σε γειτονικέ χώρες είναι μετακινήσεις. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία του προϋπολογισμού μας, είπατε. Προετοιμάζεται το Global Compact Migration για το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο πλούσια οικονομική ζώνη του κόσμου και υποδέχεται στην επικράτειά της 2,7 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες, δηλαδή λιγότερους από ότι η Τουρκία. Και εξακολουθούμε να ζητάμε από τις χώρες να κάνουν περισσότερα, αυτές που ήδη δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες. Δικαίως μας λέτε, ναι, η μετανάστευση γίνεται και συνεχίζεται τακτικά, αλλά... Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού είναι αυτή η τακτική δηλαδή μετανάστες και πού είναι οι παράνομη μετανάστες. Θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα μας στους πρόσφυγες και στις χώρες που δέχονται τους περισσότερους. Τι θα κάνουμε δηλαδή τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια γιατί εφόσον δεν υπάρχει πλέον δημοσιονομική ευελιξία εάν έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις, τις ε, που έχουμε κάνει και αν δείτε καλά για τις προτάσεις για το επόμενο πολιετές Βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βουλιάζει στους ε, εθνικούς εγωισμούς και ότι δεν έχουμε μια γενική πολιτική όπως υποτίθεται ότι έχουμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχω εξοργιστεί. Βρίσκω ότι αυτά τα δύο έγγραφα, αν τα βάλει κανείς το ένα δίπλα άλλο, σήμερα είναι πραγματικά απίστευτα σε σχέση με τις πολιτικές που κάνουμε για τους πρόσφυγες. Alors, Monsieur Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση ε, για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε σωστά τα μέσα αυτά και διαπιστώσαμε παραδείγματο χάρη πως και η πατερμοστία του για τους πρόσφυγες εν το μέσο της κρίσης δεν είχε επαρκή κονδύλια. Δεν περιμέναμε αυτά τα νούμερα και συνεργάστηκαν οι δομές ε, αλλά Βεβαίω, αυτό δεν λειτουργήσε γιατί εν μέσω κρίσεως έπρεπε διεθνείς οργανισμοί να βγουν με το καπέλο αναχείρα να ζητιανεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό η αναπτυξιακή πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών ε, έχει πραγματικά εδώ και 50 χρόνια ε, επιτύχει ή μήπως ε, έχουμε λάθος προτεραιότητες. Το θέμα επιδότηση υπερπολογισμών ή υποστήριξη έργων. Αλλά οι κατηγορίες σήμερα δεν θα μας βοηθήσουν. Το ερώτημα που πλανάτε στην αίθουσα είναι το εξής. Το θέμα είναι αν ε, τα άρθρα 78-80 της συνθήκης ε, πως δεν τηρούνται αρκετά. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Εάν ακούσουμε τα όσα είπαν οι ομιλητές και κοιτάξω τα τρέχοντα νούμερα, βλέπουμε ότι παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, όσον αφορά τις αιτήσει ασύλου, ανά μήνα, Είμαστε κάπου μεταξύ 15 και 20.000 ανά μήνα. Και στην κορύφωση της κρίσης είχαμε ε, γύρω σε 60.000 ανά μήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι εξελίσσεται. Είτε υπάρχει μία μειωμένη πίεση ε, σε αυτούς ε, οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους ή ε, κάπως απέδωσε αυτό το οποίο γίνεται με τα ταμεία στα οποία ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί στην αρχή γιατί κάτι εκτός του Κοινοβουλίου που δεν μπορεί ποτέ να το αποδεχτεί το Κοινοβούλιο αλλά φαίνεται ότι είχαμε θετικές εξελίξεις ε, στην συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε για το ποια τάξη μεγέθους μιλάμε. Ο Σφεχόφσκι ανέφερε τα νούμερα του μέσου για την, Αφρική, μια για την Τουρκία. Μια χώρα η οποία έχει κάνει περισσότερα για τους πρόσφυγες από ότι οι περισσότερες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι γίνεται επίσης με την Ιορδανία και τον Λίβανο. Δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό. Ε, Βεβαίω, ναι, εντάξει, μιλάμε για Συρία, Λιβύη και κάποιες αφρικανικές ε, χώρες. Μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποια διάσταση πηγαίνει ο κόσμος στην Τουρκία ακριβώς για να δούμε το πώς αντιμετωπίζουμε την ε, κρίση ε, για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον ε, κόσμο για να έχει δυνατότητες να παραμείνει, για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και το τι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ε, έτσι ώστε αυτή η στήριξη αν πάει τόσο θετικά όσο θέλουμε να μην αναγκάζονται να φύγουν. Αυτές ε, είναι λοιπόν οι ερωτήσεις και πώς αξιολογείτε εσείς ε, την κατάσταση εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι Πολλές φορές πήγα στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη και είχα την αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν προβάλλεται αρκετά. Συχνά περνάμε από τους διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ. Η Ευρώπη αυτή καθεαυτή δεν φαίνεται να είναι εταίρος στις χώρες όπου παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι μοιραίο αυτό ή είναι επιλογή. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά το συντονισμό. Στις διάφορες αυτές χώρες η Ευρώπη εκπροσωπείται από την αντιπροσωπεία της εκεί, αλλά υπάρχουν και αντιπροσωπείες των διάφορων χωρών και μου έτυχε να αναρωτηθώ τι επίπεδο συντονισμού υπάρχει μεταξύ των δύο. Δηλαδή η προσέγγιση μας είναι αρκετά συντονισμένη. Έπειτα, ο χάρτης πορείας που έχουν οι αντιπρόσωποι μας σε αυτές τις χώρες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χάρτης πορείας αρκετά ξεκάθαρος. Είμαστε εκεί οι παρόντες, ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί αλλά χωρίς συντονισμό, με διαδικασίες, με προθεσμίες. Κάθε φορά πρέπει τα πράγματα να φτάσουν στις Βρυξέλλες, να πούν οι Βρυξέλλες στη γνώμη τους. Υπάρχει κάποια δράνεια και κάποια δυσκολία να αντιδράσουμε έγκαιρα. Τρίτον, ακριβώς για τις διαδικασίες αυτές και πόσο βαριές είναι. Ε, το ακούσαμε ε, σε συνάντηση του Steering Board. Είναι πάρα πολλοί παρόντες, όλες οι χώρες μέλη εκπροσωπούνται εκεί και είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει τρόπο στη διακυβέρνηση να βρούμε άλλες μορφές που να μας επιτρέπουν ε, να μπορούμε να δράσουμε πιο εύκολα, να μην είναι τόσο επίσημα και τυπικά τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει μια τέτοια συνάντηση. αναρωτιέμαι η προστιθέμενη αξία που βρίσκεται σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν ευαισθησίε των μεν και των δε που θέλουμε να καλύψουμε και να καθησυχάσουμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να βρούμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς και όχι τόσο άκαμπτους. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω και οι ερωτήσεις μου κυρίως για τη διακυβέρνηση δηλαδή. Μπορούμε να παρέμβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας την εντολή από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς να ε, ηρεμήσουμε κάπως αυτήν την ε, μεταναστευτική ροή που έχουμε. Η οδύση αυτή του σκάφου του Aquarius ίσως να λειτουργήσει σαν ηλεκτροσόκ για όλους μας και να μας επιτρέψει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο πιο αποφασιστικά και πιο αποτελεσματικά. Δεν ξέρω. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ο Προεδρεύων. Άλλος κανείς. Υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις, οπότε τρία λεπτό καθένας και αρχίζουμε ανάποδα από τον κύριο Ποπόφσκι πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά λέτε. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Άντε, 3,5. Επειδή δεν χρησιμοποίησατε όλο σας το χρόνο πριν. Εντάξει, να το μοιραστώ αυτό το χρόνο με τους συναδέλφους. Λοιπόν, ναι, θα προσπαθήσω να συνδυάσω τις απαντήσεις. Θα αρχίσω με τις ειδικέ ερωτήσεις που κάνατε για την Ιορδανία, το Λίβανο, για την εκπαίδευση. Οι πληροφορίες υπάρχουν. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αναπτύξω, όλα. έδωσα παραδείγματα, το ποσοστό δηλαδή που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο στην Τουρκία, ε, και στο Λίβανο και στην Ιορδανία είναι αρκετά ψηλό το ποσοστό. Εντάξει, στην Τουρκία είναι καλύτερη κατάσταση εξαιτία και των υποδομών και ολόκληρου του συστήματος το οποίο λειτουργεί. Δεν θα σας πω όλα τα νούμερα ένα-ένα, έτσι κι υπάρχουν στην ιστοσελίδα όλα αυτά. Αλλά αν θέλετε μπορώ να τα στείλω στο γραφείο σας, ώστε να τα έχετε. Το μοντέλο είναι λίγο πολύ το ίδιο. Χτίζονται σχολεία, υλικό σχολικό, κατάρτιση δασκάλων, στην Τουρκία κυρίως γλωσσική εκπαίδευση. Ε, προσλαμβάνονται επίσης δάσκαλοι στη, στο Λίβανο και στην Ιορδανία επειδή ακριβώς οι κοινότητες προσφύγων είναι τεράστιες. Έπειτα, ρωτάτε για την μεταναστευτική πίεση στην πηγή. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η δράση μας έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς. Αν δούμε τι γίνεται στην κεντρική Μεσόγειο, η σύγκριση των περσινών στοιχείων του 17 δηλαδή με το 16 είναι 47% λιγότερες αφήξεις. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πίεση, εξακολουθεί να υπάρχει ο κόσμος, εξακολουθεί να φεύγει και να θέλει να έρχεται σε μας αλλά λέω ότι υπάρχει πάντως μείωση του ποσοστού. Σίγουρα χρειάζονται προσαρμογές, το παραδέχομαι. Στο επόμενο στάδιο για την διευκόλυνση με την Τουρκία πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την εκπαίδευση, την υγεία, αλλά και στην απασχόληση πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κοινοτικό επίπεδο. Και αυτό θα είναι στοιχείο κλειδί τα επόμενα χρόνια. Τέλος, όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση και την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, συμφωνώ. Είναι πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη, στους στόχους δηλαδή του Επιτρόπου Χαν. Όντως, θέλουμε να είμαστε ορατοί. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που κάνουμε ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε εμείς που τα κάνουμε. Σίγουρα οι διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ κάνουν τεράστια δουλειά. Το 40% πηγαίνει μέσα από διεθνείς ε, οργανώσεις, κυρίως ε, του ΟΗΕ, UNICEF ε, και άλλες. Δεν λέω ότι θα αλλάξει αυτό. Αλλά είμαστε προσεκτικοί και έχουμε διάλογο μαζί τους. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο υλοποιούνται όλα αυτά. Ξέρω ότι κάποια από αυτά τα σώματα είναι τεράστια. Οι χώρες μέλη, είναι αλήθεια, ότι δίνουν μεγάλη σημασία στη Steering Committee όσον αφορά τη διευκόλυνση για την Τουρκία. Και από νομική άποψη αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το κάτι καταπιστευματικό ταμείο. Όλες οι χώρες μέλη συνεισφέρουν γι' αυτό και έχουν μια έδρα εκεί. Αν πάρουμε όμως το καταπιστευματικό ταμείο για την ε, Συρία, είναι πολύ πιο μικρό. Γιατί θα πρέπει να είναι ένα δισεκατομμύριο Ό,τι είναι λιγότερο δεν ε, εκπροσωπείται. Οπότε έχουμε ένα, μια μικρότερη ομάδα. Έτσι έχει. Τι να κάνουμε για λόγους ε, λογιστικούς, διαφάνειας. Έτσι είναι. Ελπίζω πάντως να ε, μπορούμε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και πολύ χαίρομαι που μας δίνετε ευκαιρία να ακούσουμε και τη γνώμη σας εδώ και τις ιδέες σας. Παρακαλώ, Κύριο Ντούς. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω για την ειλικρίνεια των αποτελεσμάτων. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε για τα αποτελέσματα είναι, και διαβάζω εδώ, εξωτερική δράση είναι ακριβώς επειδή έχουμε την τάση να παρουσιάζουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι πάντα καλύτερα κάποιος να σας λέει ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο από ότι είναι μισοάδιο, σωστά. Πάντως δεν έχουμε βρει το μαγικό ραβδί που θα μας επιτρέψει να αφαιρέσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη. Αν δω ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, το, η κλιματική αλλαγή, είναι κάτι που μόνο πρόσφατα έχει αρχίσει να μπαίνει στο κάδρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αρχίσουμε πάντως να βλέπουμε αποτελέσματα επιτόπου. Βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που δοκιμάζουμε και σε αυτά που λειτουργούν, με αυτά που δοκιμάζουμε και δεν λειτουργούν. Πολύ σημαντικό αυτό σαν ε, μέσω Τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί επί τόπου. Η ίδια προσέγγιση με αποχρώσεις πρέπει να εφαρμοστεί και στις πολιτικές. Λέτε τι δυσκολίες που είχαμε με τη δήλωση της Βαλέτα, με τη δήλωση του Αμπιτζάν επίσης. Είναι αλήθεια ότι όταν έχουμε μια καθαρά πολιτική συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο, έχουμε την τάση να συζητούμε για αρχές πυλώνες, ισορροπίες. Είναι δύσκολο. Τώρα όμως που δραστηριοποιούμεθα επί τόπου, είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχουμε συγκλήσεις με τους εταίρους μας. Δηλαδή, ποια είναι η δράση αυτή που καλά θα κάνουμε να χρηματοδοτήσουμε και ποια καλά θα κάνουμε να μην χρηματοδοτήσουμε. Βλέπουμε δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει τους εταίρους μας να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν, που είναι δικές τους, δεν δικές μας, έτσι. Εδώ μπορεί εύκολα να επιτευχθεί σύγκληση. Και έτσι φτάνω και στη διακυβέρνηση, το Συμβούλιο και οι διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι τέτοιες συναντήσεις μεγάλες φαίνονται έτσι πολύ βαριές και άκαμπτες. Όμως το Στρατηγικό Συμβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό φόρουμ συνάντησης. Εκείνη που γίνεται η συζήτηση για τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που θέλουμε να ακολουθήσουμε με το καταπιστευματικό ταμείο. Γι' αυτό και γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που δεν κάνουμε στο επόμενο επιχειρηματικό πλαίσιο, επιχειρησιακό μάλλον πλαίσιο. Για το συντονισμό με τις χώρες μέλη τώρα, γίνεται. Όπως πάντα οι χώρες μέλη είναι πιο πρόθυμες να μας συντονίζουν εμάς παρά να τις συντονίζουμε εμείς. Πάντως, ό,τι κάνουμε με τα καταστηματικά ταμεία συζητιέται και στην κάθε χώρα και γίνεται συντονισμός των δωρητών ώστε να δούμε τι κάνουν και άλλες πλευρές στην κάθε χώρα. Γίνεται συντονισμός λοιπόν με τις χώρες μέλη και λειτουργεί μάλλον καλά. Και αυτό εξηγεί γιατί μετά όταν αρχίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις για συγκεκριμένα προγράμματα, συνήθως τα πράγματα πηγαίνουν εύκολα, γιατί ακριβώς η προπαρασκευαστική δουλειά έχει ήδη γίνει στην αρχή. Τέλος, όσον αφορά την προβολή του έργου μας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Συχνά όμως, εκτός βέβαια όταν περνάμε από ε, τις υπηρεσίες του ΙΕ, είναι κάτι που είναι γνωστό από τους εταίρους μας και από τους τελικούς δικαιούχους. Από πού δηλαδή προέρχονται τα χρήματα. Ε, ποιος ασχολείται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις τοπικές ε, αρχές, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται. Μερικές φορές η προβολή είναι πολιτική και δεν συνδέεται απαραίτητα με την ευρωπαϊκή σημαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριο. Λεφλέρ. Ευχαριστώ, είπαν ήδη αρκετά οι δύο συνάδελφοι. Εγώ θα προσθέσω απλά κάποια στοιχεία. Θα ξεκινήσω με τις διάσημες ε, αιτίες ή πηγές. Ε. ε, όπως το είπατε κύριε Πρόεδρε, πώς θα... Μπορέσουμε να σταματήσουμε τις πηγές της μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ούτε και θέλουμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε να παρέμβουμε για να σταματήσει η αναγκαστική ε, μετακίνηση αλλά η μετανάστευση, η ίδια η μετανάστευση, κατά τη γνώμη μου, είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος ανέκαθεν μετακινούνταν, ανέκαθεν έψαχνε νέους ορίζοντες. Το, το δικό, η δική μας πρόκληση είναι να πλαισιώσουμε τη μετανάστευση, να την καταστήσουμε επιλογή και όχι ανάγκη και αυτό εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα της διαθετικής μας βοήθειας στις προσπάθειες που κάνουμε μακροπρόθεσμα με τους εταίρους μας στην Αφρική, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί ε, ακριβώς προσπαθούμε να ε, βρούμε γενικές αναφορές που περιλαμβάνουν διάφορες διαστάσεις, διακυβέρνηση, κοινωνική. Κοιτάξτε, όταν είπα ότι πρέπει να σταματήσουμε τις πηγές, ναι, η μετανάστευση είναι το ίδιο αρχαία όσο και η παγκοσμιοποίηση. Μπορεί όμω να είναι τέτοια τα φαινόμενα που να επιταχύνεται η διαδικασία και να δίνονται λόγοι για μετανάστευση και σε κόσμο που αρχικά θα προτιμούσε να μείνει σπίτι του. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά όπως είπε και η κυρία Κολέτε, συχνά είχαμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο όπου όταν περνάμε από την υποανάπτυξη προς μία ανάπτυξη, αλλά είμαστε ακόμα σε μια φάση αρχική, συχνά υπάρχει μια επιτάχυση της μετανάστευσης γιατί οι άνθρωποι έχουν περισσότερα μέσα ενώ έχουν προσδοκίες οι οποίες, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται δεν πραγματοποιούνται γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να, βρουν μια ικανοποίηση, να μπορούν να έχουν ένα μέλλον εφόσον το αναζητούν και αν το επιθυμούν στη δική τους κοινωνία και κοινότητα. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θέλουν να, να πάνε αλλού, όπως το έχουν κάνει και εκατομμύρια εκατομμυρίων Ευρωπαίοι. Εδώ μιλάμε για πλαισίωση της νόμιμης μετανάστευσης. Γι' αυτό και γίνονται οι διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του ΟΗΕ για το παγκόσμιο σύμφωνο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διαπραγματεύσεις για να έχουμε ε, αναγνώριση της κοινή ευθύνη όλων, όλης της διεθνούς κοινότητας. Η Λίντα Μακάβαν ρώτησε για την διάρθρωση μεταξύ των εξωτερικών μέσων και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών η απάντηση είναι ότι τα εσωτερικά μέσα εστιάζουν κυρίως το τι κάνουμε εντός της Ένωσης για να διαχειριστούμε την μετανάστευση και όσον αφορά την δυνατότητα υποδοχής και δυνατότητα ελέγχου συνόρων κτλ. Θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε στην εξωτερική ε, διάσταση ε, όχι να έχουμε ένα ξεχωριστό μέσο μετανάστευσης, αλλά να είναι ένα από τα βασικά σημεία. Κυρίως και επίσης γιατί υπάρχει τόσο πολύ μετανάστευση μεταξύ άλλων υπήρων και άλλων χώρων. Και εγώ ε, ήμουν πρόσφατα σε έναν τέτοιο διάλογο με την Νότια Αφρική και είναι εκπληκτικό το πόσο παρόμοιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Νότια Αφρική. Ε, με κάποια κράτη-μέλη και πόσο ακριβώς θέλουν να μοιραστούν εμπειρίες. Ακριβώς για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα και τις ξενοφοβίες και τα λοιπά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα που πρέπει να δούμε ε, και πρέπει να τα δούμε ελπίζω με μεγαλύτερη ευελιξία με τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές για να συνδυάσουμε ακριβώς εσωτερικές και εξωτερικές ε, πτυχές. Όπως ανέφερα, παραδείγματος χάρη ε, και με το θέμα του Αμπιτζάν, με την Αφρικανική Ένωση, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη υιοθέτηση και ενδιαφέρον. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. συμφωνώ ότι ε, είναι ε, εντυπωσιακό το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως είπε και η Λίντα Μακάβεν πρέπει ακριβώς να δώσουμε βάρος στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε έναν πραγματικό στρατηγικό σχεδιασμό ε, εμπλέκοντας και το Κοινοβούλιο ε, πέρα από τις καθαρά τεχνικές πτυχές των έργων που βλέπουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κολέτ. Για μια πολύ σύντομη παρέμβαση παρακαλώ. Κοιτάξτε, ακούστηκαν τόσα πολλά. Οπότε θα περιοριστώ σε ε, κάτι το τελευταίο. Υπάρχει μια προειδοποίηση και μια ευκαιρία. Πρέπει να αποφύγουμε την ύβερη, δηλαδή το τι μπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια όρια. Και το τι θέλει να επιτύχει, εντάξει, να μιλάμε για διαχείριση συνόρων και εξωτερικοποίηση κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχει μια συζήτηση ανάπτυξη και για τι αιτίε. Η πολυπλοκότητα αυτή τη δυναμική είναι τεράστια. Και βεβαίω τώρα υπάρχει πίεση για να μπει ως πρώτη προτεραιότητα η μετανάστευση. Και ακριβώς τώρα το θέμα είναι να δούμε πού ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε τη μετανάστευση στον προϋπολογισμό, ποιοι στόχους θέλουμε να επιτύχουμε και πώς ελαχιστοποιούμε τις συγκρούσεις των ενδιαφέρων στόχων και χαρτοφυλακίων που ακόμα νομίζω βρίσκονται σε μια διαδικασία συμβιβασμού, δηλαδή ανάπτυξη, ανθρωπιστικά και τα λοιπά. Οπότε τώρα υπάρχει νομίζω μια ευκαιρία ακριβώς να σκεφτούμε εις ε, το θέμα αυτό. Να δούμε δηλαδή πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε ε, αποτελεσματικά και ποιος θα τα υλοποιήσει. Ευχαριστούμε πολύ τους τέσσερις εμπειρογνώμονες. Τώρα, η πρόεδρος της ΔΕΒΕ πρέπει να έρθει εδώ. Και αντιπρόεδρος Κόντου. Καλησπέρα συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Όπως βλέπετε έχουμε δύο νέους συμπροέδρους, ε, εμένα, ε, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και την συνάδελφο, την κυρία Λίντα Μάκαβαν, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης. Δύο Βρετανούς δηλαδή, συμπροέδρους, τη εργαζόμαστε σκληρά, μήπως και φύγουμε σε νέα μήνες. Τέλος θα δούμε. Είναι το πρώτο πάνελ, ε, λοιπόν. Υπάρχει νομίζω αρκετά μεγάλη άλλη επικάλυψη ε, όπως ε, τα είχαμε δει και στο πρώτο πάνελ για το τι συμβαίνει αυτήν την στιγμή και να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο αντίκτυπος των δράσεων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω επιπρόσθετων ή νέων ειδών χρηματοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι ε, μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα γιατί υπάρχει και απάτη και διαφθορά με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την αποτελεσματικότητα βεβαίως αν υπάρχουν αποτελέσματα τελικά επιτόπου. Οπότε αυτά είναι εξίσου σημαντικά. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε αυτό το εργαστήριο σήμερα το απόγευμα για να δούμε τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι έχουμε τέσσερι ειδικού ε, εδώ πέρα για να μα ε, εκφράσουν την άποψή του. Τον κύριο Μασούντου, Υπουργό Οικονομικών του Νίγηρα, ο κύριος ε, Μπιερή από την Κονκόρντο, την Ένωση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ε, ΜΚΟ Αναπτυξιακής Συνεργασίας και την ε, κυρία εδώ, η οποία είναι ειδική στην μετανάστευση, ο κύριος Γιούρεκ από το Βρετανικό Συμβούλιο και ασχολείται συγκεκριμένα με την αναπτυξιακή συνεργασία και ο Μπομπάρνολ επίσης από το Βρετανικό Συμβούλιο, ο οποίος ε, διευθύνει το Αναπτυξιακό Τομείο της Νιγηρίας ε, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπω ο τίτλος σας είναι πολύ μακροσκελής. Οπότε προχωράμε και σας δίνω τον λόγο. Δίνω τον λόγο στην αγαπητή συμπρόεδρο Λίντα. Ευχαριστώ Τέρεκ. Ε, ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους. Ε, έχουμε ένα από τα πιο ε, πιεστικά ζητήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές, χαίρομαι που έχουμε τον Υπουργό εδώ από τον Νίγηρα Και βεβαίως ε, εγώ ανήκω στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σας είχε επισκεφθεί ο πρόεδρός μας, ο Κλοντ Μωραές, ε, είχε επισκεφθεί τον Νίγηρε. Ε, ακριβώς για να δούμε το θέμα της χρήσης του καταπιστεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρχε και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τον κύριο Υπουργό για το πώς αξιολογεί τα ωφέλη, όπως τα βλέπετε εσείς, ε, που έχει η χώρα σας. Και, και να είμαστε και ειλικρινείς ε, βεβαίως. Ε, τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα. Πρέπει να συζητάμε τα προβλήματα όταν ήμουν στην Ουγκάντα, ε, όπως είπαμε, είχα, η Επιτροπή μας τον Μάιο, πριν από ένα μήνα, είδαμε εκεί πέρα πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Και βεβαίως οι πρόσφυγες ήταν κυρίως γυναικόπαιδα από τον Νότιο Σουδάν που περνούσαν στην Ουγκάντα και βεβαίως η αλλαγή της ε, πολιτικής ε, ήταν ότι αντί να δίνονται κονδύλια στους πρόσφυγες η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζε όλον τον πληθυσμό της περιοχής ε, που αισθάνεται ότι δεν τον βοηθάνε και θεωρούσαν ότι βοηθούσαν μόνο τους ε, πρόσφυγες και οφείλω να πω ότι όπως είπε και ένας ομιλητής ε, δεν είναι οι αφρικανικές χώρες ε, ιδιαίτερα. Ε, κυρίως οι αφρικανικές χώρες φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και όχι στην Ευρώπη παρά τα όσα δείχνουν τα δικά μας μήμη και φιλοξενεί εκεί πέρα η Ουγγάντα το μεγαλύτερο ρυθμό προσφύγων μετά την ε, Τουρκία στον κόσμο και είναι μία από τις στοχότερες χώρες στον κόσμο και θέλω να ακούσω και περισσότερα από την Concord Νομίζω ότι εκπροσωπούν ε, τις υπηρεσίες των ε, κρατών ε, μελών. Η Concord θα μας πει την πτυχή των ΜΚΟ. Και έχουμε τον Μπομπάρνολτ εδώ πέρα, ο οποίος ήρθε από την Ιγυρία για να μας πει το πώς έχουν τα πράγματα επί τόπου. Ακριβώς αυτό δεν το έκανα για να ασκήσω κριτική, αλλά να ακούσουμε και τα θετικά και τα άσχημα. Ε, υπήρχαν κάποια προγράμματα των ΜΜΕ που λέγανε ότι πού πάνε τα λεφτά, σε πιάνουν τα χέρια καταλήγουν. Ε, θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε ποιες είναι οι σχετικές προκλήσεις. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον Υπουργό Μασούντου του Νίγηρα για 8 έως 10 λεπτά. Έχετε τον λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε να παρακολουθήσω την συνεδρίασή σας. Ε, πρόκειται για θέματα που είναι πολύ ανησυχητικά για σας και για μας, ε, τα θέματα της μετανάστευσης και που σήμερα απειλούν την δημοκρατική ισορροπία των χωρών σας. Είναι πολύ μεγάλη ε, ως προβληματισμό λοιπόν για σας, αλλά και για μας. Θα ήθελα επίσης να πω κάτι που δεν είναι προφανές. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς υποδεχόμαστε ε, πρόσφυγες αλλά και επαναπατρισμένους ενώ είμαστε μια χώρα εξαιρετικά φτωχή ε, δεχτήκαμε για παράδειγμα 200.000 ε, πρόσφυγες μετά από την κρίση της Λιβύης 300.000 μετά από την κατάσταση που προκάλεσε τον Μπόκο Αράμα στο Τσάντ και στην Ιγυρία, στη Βόρεια Νιγηρία και μετά από το κρίση του Μαλή έχουμε 600.000 ε, ε, δηλαδή πρόσφυγες συνολικά για ένα πληθυσμό 20 εκατομμυρίων και σε μια χώρα εξαιρετικά φτωχή. Το ζήτημα λοιπόν ε, το προσφυγικό το ζούμε και εμείς. Προφανώς η συζήτηση που γίνεται εδώ είναι πολύ ανησυχητική για τους δικούς σας και είμαστε αλληλέγγυοι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βρεθεί λύση να συνεχίσουμε να βρούμε ε, ε, διεξόδους ώστε να είναι πάντοτε ανθρώπινες και δημοκρατικές. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα γιατί ο Νίγηρας λόγω της γεωγραφίας του ε, έτσι όπως είναι δηλαδή η γεωγραφική του θέση ξέρω το γνωρίζετε αλλά καλό είναι να σας θυμίσουμε καταρχάς είμαστε μια χώρα διέλευσης έχουμε Πρόκειται για μια χώρα που συνορεύει βόρειο-ανατολικά με την Λιβύη. Ε, συνορεύουμε λοιπόν, έχουμε κοινά σύνορα με την Λιβύη. Έχουμε επίσης χίλια χιλιόμετρα σύνορα με την Αλγερία βόρεια. Έχουμε 800 χιλιόμετρα σύνορα με το Μαλί, με το βόρειο Μαλί. Στο βορειοδυτικό μας τμήμα συνορεύουμε λοιπόν με το Μαλί, στα δυτικά με το Τσάντ και Νότια έχουμε 1500 χιλιόμετρα σύνορα με την Ιγυρία. Είμαστε δηλαδή σε ένα σταυροδρόμι της ζώνης της κρίσης. Είμαστε χώρα ε, διέλευση. Η πόλη Γκαντέζ που είναι το κεντρικό στοιχείο της διέλευσης αυτής είναι βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος. Σε σε μια ακτίνα χιλίων χιλιόμετρων γίνονται όλα αυτά, δηλαδή ανάμεσα στα Καντέζ και τα σύνορα της Λιβύης και της Μπουρκίνας και του Μαλή. Έχουμε δηλαδή ένα ε, τεράστιο χώρο που πρέπει να ελέγξουμε. Είναι λοιπόν ε, φαντασ... Ε, τεράστιος ο χώρος που πρέπει να ελέγξουμε για να συμβάλλουμε στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Να θυμίσω ότι επίσης όλα αυτά γίνονται σε μια ευαίσθητη χώρα ε, που έχει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των κλιματικών αλλαγών. Όλοι μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά σε εμά οι κλιματικές αλλαγές έχουν συγκεκριμένο πρόσωπο. Παλιότερα είχαμε μια χρονιά ξηρασίας στις 10. Ε, μετά έγινε μία στις 5 χρονιές, τώρα είναι μία στις 2 χρονιές η ξηρασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πράγμα το οποίο φτωχοποιεί τον πληθυσμό και δημιουργεί εξαιρετικά τεταμένες καταστάσεις. Επίσης, ε, στη δεκαετία 80-90 στις χώρες αυτές, στην περιοχή του Σεχέλ και στη Δυτική Αφρική γενικά, είχαμε τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν γίνεται πολλή λόγο για αυτά, αλλά είχαν ω συνέπεια διότι έπρεπε να σταματήσουν οι κοινωνικέ δαπάνε, έπρεπε να σταματήσουν οι δαπάνε για την ασφάλεια. Όλα αυτά είχαν ω ε, ε, συνέπεια, για εμά είναι τα χαμένα χρόνια, έτσι τα λέμε. 80 μέχρι άντε και 2.000. Γιατί ο κόσμος έγινε πολύ πιο ευάλωτος και αυτό ξεκινά από την περιφέρεια. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε κράτος. Και στη συνέχεια είχαμε την κρίση της Λιβύης κατά την κατάρρευση του Λιβικού κράτους που επιτάχυνε τα προβλήματα προβλήματα για την ασφάλεια στο σύνολο του Σαχέλ και δημιουργήθηκε έτσι και αυτό κενό. Το κρατικό κενό. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένας κρατικός έλεγχος, δεν υπήρχε κράτος. Φυσικά και ε, ε, ε, ήταν βάσιμοι λόγοι που προκλήθηκαν όλα αυτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση έκανε μετάσταση σε ολόκληρη τη ζώνη. Είχαμε λοιπόν ευαίσθητη κατάσταση στις περιφέρειες της χώρας και σταδιακή αλλαγή με την κατάρρευση των χωρών. Εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας. Περάσαμε από μια φυσιολογική οικονομία όπου ε, στο ζώνη Αγκαντές ο τουρισμός ήταν η βασική μας ε, ε, δραστηριότητα αλλά αντικαταστάθηκε αυτό από την εγκληματική οικονομία που χαρακτηρίζεται από δύο ειδών οικονομίες, δηλαδή ναρκωτικά και μετά από την κατάρρευση των κρατών, από τις γύρω-γύρω κρατών και ε, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και λαθρεμπόριο των προσφύγων αφού κατέρευσε η Λιβύη. Αυτό αυτή η εγκληματικού τύπου οικονομία αναπτύχθηκε πολύ, άνθησε πολύ και πολλοί κόσμος αυτές τις ζώνες ζει άμεσα ή έμεσα από αυτές τις εγκληματικές οικονομίες και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και προσφύγων ή μεταναστών. Δεν πρέπει να βλέπουμε το πράγμα δηλαδή μόνο και μόνο ε, λες και είναι κάτι το οποίο είναι ε, γηγενές πρόκειται για την οικονομία ολόκληρων περιοχών, ολόκληρων πληθυσμών που πρώτα ζούσαν από τον τουρισμό και τώρα ζουν βασικά από αυτή την οικονομία. Άρα λοιπόν για μας είναι μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια θέμα ασφάλειας, κάναμε πολλά πράγματα και είχαμε αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Και ακόμα και βραχυπρόθεσμα είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Σας είπα ότι έχουμε μία ακτίνα χίλιων χιλιόμετρων. Πώς να ελέγξουμε όλο αυτό το χώρο με τόσο περιορισμένα μέσα. Εκτιμούμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ε, δυνάμεις ασφαλείας μας. Δημιουργήσαμε και ένα ειδικό αστυνομικό σώμα, αλλά είναι τεράστια τα μέρη. Ε, ε, είχαμε παρόλα αυτά ε, σημαντικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον έλεγχο των ροών που περνούν από τον ε, Νίγηρα. Αλλά δεν είναι βιώσιμο αυτό, δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ, για πάντα. Πώς θα ε, αντικαταστήσουμε την παράνομη οικονομία από μια νόμιμη που θα επιτρέψει να μην χρειάζεται η παράνομη οικονομία. Αυτό είναι το, βασικό θέμα. Και έπειτα πρέπει οπωσδήποτε, επειδή είδαμε ότι αυτό είναι το βασικό αίτιο, η κατάρρευση των κρατών ή εν πάση περιπτώσει η αποδυνάμιση των κρατών, πώς θα αποκατασταθεί το κράτος στις ε, βασικές του δραστηριότητες και αρμοδιότητες. Έπειτα, επιστροφή της διοίκησης, μόνιμη παρουσία της διοίκησης ε, των ε, της αστυνομίας αλλά και των βασικών ε, ε, εργασιών του κράτους, δηλαδή νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Ε, υπάρχουν δηλαδή ανάγκες επίγουσες. Πρέπει να σκεφτούμε όμως και τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, ε, να αντικατασταθεί με βιώσιμο τρόπο η εγκληματική οικονομία από μια φυσιολογική οικονομία και δεύτερον να αποκατασταθεί το κράτος στις κοινωνικές του λειτουργίες και στις ε, δικαιωτικές του λειτουργίες. Και αυτό απαιτεί πολλούς πόρους και δεν είναι χαμένα λεφτά. Και γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική έλεγχο, δημοσιονομικός έλεγχος και ανάπτυξη αλλά και συντονισμός όλων αυτών των δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των κρατών γιατί αλλιώς απαξιώνεται το κράτος. Αυτά εν ολίγης και σύντομα για το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Όντω υπογραμμίσατε τα ζητήματα έτσι όπως τα βλέπετε εσείς από την πλευρά σας. Ε, ο ρόλος σας είναι τεράστιος βέβαια, δεδομένου ότι ζείτε σε μια περιοχή γύρω-γύρω από την οποία βρίσκονται ασταθείς ε, χώρες ή καθεστώτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για αυτά που μας είπατε. Τώρα η Φάνη Μπιχάρη έχει το λόγο από την Concord. Δεν ξέρω από ποιο τμήμα της Κονκόρτ ακριβώς προέρχεστε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα και μιλάω μετά τον κύριο Μασαντού. Θα σας πω λίγα πράγματα για την ανάγκη χρηματοδότησης ε, της μετανάστευσης. Είμαι μέλος της Act Alliance EU Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών. Ο σεβασμό ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία τη ισότητα, του κράτου δικαίου και ο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, απαγορεύεται η μαζική απέλαση, κατά το οποίο σημαίνει επίση ότι υπάρχει και η μη επαναπροώθηση. Όλα τα κρατημέλη έχουν υπογράψει την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κατά το οποίο δεσμεύει και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Μέσω του μέσου χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει τον σεβασμό των αξιών στα κράτη-μέλη και χάρη στον προϋπολογισμό εξωτερικής δράσης μπορεί να ενισχύσει αυτές τις δράσεις και σε υποψήφιες χώρες. Όμως, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά τα χρηματοδοτικά για να ασκήσει πίεση σε τρίτες χώρες και να επιδιώξει τα δικά τη συμφέροντα με το να θέσει όρου ε, που θα αφορούν την ευθυγράμμιση με τις προσδοκίε τη ω αποτέλεσμα της ε, μεταναστευτική ε, κρίσης έγιναν σημαντικέ αλλαγέ στα χρηματοδοτικά μέσα για την εξωτερική δράση. Η προσπάθεια της Ένωσης να μειώσει την μετανάστευση βασίζεται στην συνεργασία με τρίτες χώρες, ε, την αντιπροσωπευτικότητα των αρχών της ανάπτυξης και την εξάλληψη της φτώχειας. Ένα παράδειγμα είναι το καταπίστευμα για την Αφρική, όπου υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και πολλά παραδείγματα αρνητικής επίδρασης ε, στην περιφερειακή ικανότητα, στην οποία βασίζεται το βιός των ανθρώπων. Δεν υπάρχει συνεργασία με τις χώρες οι οποίες λαμβάνουν τη χρηματοδότηση ε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Η εργαλειοποίηση της βοήθειας αυτής για τα συμφέροντα επίπεδου εξωτερικών ε, πλέον σημαίνει ότι η μετανάστευση θα παραμείνει στην πολιτική ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς οι μετανάστες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε κάποια προγράμματα. Εντάξει, όσο αναγκαίο και αν είναι, η ευελιξία και τα προγράμματα τα οποία μόνο γύρω από τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, επίσης, ε, έχει τον κεντρικό ρόλο στον προϋπολογισμό. Δεν γίνεται έτσι να ενισχυθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, ούτε ένα τρόπος ελέγχου της μετανάστευση προς την Ένωση. Οι κοντόφθαλμες λύσεις ε, που ακολουθούν κάποια αμφιλεγόμενα προηγούμενα, όπως η συμφωνία με την ε, Τουρκία ή με την Λιβύη, που διακινδυνεύουν ζωές, αγνοούν και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ρόλος ε, αλλά θα πρέπει να ξοδεύουμε χρήματα στις χώρες τέρους ε, και να υπάρχουν κάποιες τακτικές ε, δίωδοι και για να ευνοηθούν και οι χώρες που εξαρτώνται από την μετανάστευση για την ανάπτυξή τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν κάποιοι τρόποι οι οποίοι θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχουν αξιοπρέπεια και επίσης να σεβόμαστε την αρχή της μη επαναπροώθησης και την απαγόρευση συλλογικών απελάσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιείται αναπτυξιακή βοήθεια για καταναγκαστικές επιστροφές. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τις αιτίε ε, αυτές, αλλά πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο, σε συνεννόηση με τους μετανάστες, ε, τις κοινότητες που φιλοξενούν και τις τοπικές κυβερνήσεις. ανάγκες γυναικών, παιδιών και παθών ομάδων επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο στόχο της χρηματοδοτική στήριξης θα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν βιώσιμε λύσει που θα αντιμετωπίζουν ε, τις ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές διαδικασίες, το κράτο δικαίου, την δικαιοσύνη των φίλων και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, όχι να σταματήσουν τη μετανάστευση. Η συνεργασία με χώρε που φιλοξενούν εκτοπισμένου πληθυσμού θα πρέπει επίσης να έχει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική δράση, καθώς πάνω από 80% των εκτοπισμένων παραμένουν σε αναψώμενες χώρες. Οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο εάν οι ντόπιοι εκπρόσωποι και οι ντόπιες κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με τρόπο ουσιαστικό στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων. Επίση θα πρέπει να στηρίξουμε και τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Όλοι αυτοί οι τομεί θα πρέπει να συνοδευτούν από προγράμματα που θα στηρίζουν τα άτομα που χρήζουν διεθνού ε, προστασία. Για να διασφαλιστεί η μη επαναπροώθηση και το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και βεβαίω επειδή είναι ο πρώτο δότη ε, παγκοσμίω στο τωρινό πολιτικό κλίμα έχει μεγάλη σημασία να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών. Και αναμένουμε την συνεργασία μαζί σα ε, στις λεπτομέρειες του επόμενου προπολογισμού. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ και περνάμε τώρα στους δύο τελευταίους ομιλητές. Έχουμε τον Κρις Γιούρικ, που είναι διευθυντής ε, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξική Συνεργασία και τον Bob Arnott, που είναι διευθυντής του Trust Fund για την Βορειοανατολική Νιγερία. Παρακαλώ, ο κύριος Γιούρεκ πρώτα. Ευχαριστώ. Όντω είμαι εκπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Εδώ σε τρία λεπτά θα σας πω οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα επιτόπου τι κάνουν και θα δώσουμε και κάποιες προοπτικές όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων. Λοιπόν, είμαστε ένα δίκτυο 15 ευρωπαϊκών ε, οργανώσεων και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έρθει και η λιθουανική αντίστοιχη οργάνωση που θα συμπληρώσει το δίκτυο. Θέλουμε να μοιραστούμε πραγματογνωμοσύνη μεταξύ μας και να βελτιώσουμε ε, το πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό. Οπότε ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ. Ελπίζω να μπορούμε να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας ώστε να διευκρινίζουμε και τα πράγματα. Το δίκτυο αυτό φροντίζει την αποκοινού υλοποίηση μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, ώστε να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα. Και τώρα έρχομαι στο Καταπιστευματικό Ταμείο Επίγουσας Βοήθειας. Οι περισσότεροι στο δίκτυο δουλεύουν μέσω καταπιστευματικού ταμείου και μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικοί τρόποι για να γίνει αυτό, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινέ τάσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Συνένεση και όντως έχει επιτευχθεί αυτό για να πετύχουμε και τις δεσμεύσεις για το 2030. Όσον αφορά τη διαφάνεια, αναγνωρίζουμε από την αρχή ότι οι αποφάσεις και η χρηματοδότηση επιδέχονται βελτίωση, όπως επίσης η διαφάνεια, γιατί πρέπει να είναι δημόσια όλα αυτά και να διέπονται από πλήρη διαφάνεια. Τα καταπιστευτικά ταμεία προσφέρουν βέβαια μια πολιτική δέσμευση και δρούν καταλυτικά για τη συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά τη μετανάστευση και ε, ρίχνουν τους προβολείς ε, πράγματι σε κάποιες ομάδες που αλλιώς ε, δεν εμφανίζονται καθόλου. Θέλουμε να βοηθήσουμε βέβαια τη δικτύωση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό γίνεται μέσω των καταπιστευματικών ταμείων. Οπότε η προσδεδεμένη αξία των ταμείων αυτών προσφέρεται ακριβώς εκεί που δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, με ευελιξία, διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλα αναπτυξιακά μέσα. Το δίκτυο όμως πιστεύει ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του καταπιστευματικού αυτού ταμείου επίγουσας βοήθειας είναι ότι δίνει γρήγορα λύσεις μέσα σε ένα απλό ε, σε μια απλή δομή λήψης αποφάσεων. Και προσφέρει επίσης και από κοινού υλοποίηση λύσεων με μεγαλύτερη ικανότητα και με πιο εύκολα πλαίσια που δρούν επιτόπου. Επίσης υπάρχει μεγάλη προσαρμοστικότητα στην υλοποίηση. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση επιτόπου κάθε φορά και να υπάρχει και ενστερνισμός από την τοπική κοινότητα. Ακόμα και αν οι δομέ των εταίρων μα επιτόπου είναι πολύ αδύναμε. Επίση, το Καταπιστευματικό Ταμείο προσφέρει καλύτερη συνεργασία και συντονισμό των δωρητών με συντονισμένη προσέγγιση που βασίζεται στα στοιχεία που έχουμε από το Καταπιστευματικό Ταμείο Επίγουσας Βοήθειας. Όμως αναγνωρίζουν τα μέλη μας ότι μερικές φορές υπάρχουν υπερβολικά πολλά στρώματα που εμποδίζουν την διαφάνεια της παρέμβασης. Σίγουρα χρειάζεται και περισσότερη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη επιτάχυνση της αντίδρασης όταν υπάρχει Επιγούς ανάγκη. Συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει τις διευκολύνσεις σε όλους όσους δρούν επιτόπου και να ληφθούν υπόψη πραγματικότητες επιτόπου. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Μποπ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ από την πλευρά μου. Στην Ιγυρία δουλεύω τα τελευταία 15 χρόνια Έχω ένα κατεπισμαστικό ταμείο πρόγραμμα. Ε, εμείς είμαστε στον Πόρνο και αλλού, όπου δράει και τον Πόκο Χαράμ. Έχουμε 30 διαφορετικές κυβερνήσεις με τις οποίες είμαστε σε επαφή. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό πέρα από τις ερωτήσεις που θα προσπαθήσω να απαντήσω που υπάρχουν στο έγγραφο αλλά θα σας πω κυρίως τι αντιμετωπίζουμε εμείς όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω, που υπόθηκε ήδη σε υψηλό επίπεδο, είναι το θέμα της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας. Αυτό το οποίο εμείς ζητούμε από το καταπιστευματικό ταμείο για τα προγράμματά μας είναι αυτό. Κυρίως στα πλαίσια μέσα στο οποίο δουλεύουμε, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια ευκαιρία πρέπει να είμαστε θέση να τη δράξουμε. Και αντίθετα, κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να μπορούμε να αποσυρθούμε. Είτε πρόκειται για δυσκολίες ε, καθαρά φυσικές. Πρέπει λοιπόν το πρόγραμμα να είναι ευέλικτο κάθε φορά και να προσαρμόζεται στις επιτόπου συνθήκες. Αυτή είναι μια έκκληση που κάνουμε λοιπόν για τα προγράμματα. Πρέπει να υπάρχει προσαρμοστικότητα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Το δεύτερο που θα λέγαμε είναι ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ε, που να μας βοηθάει να αποφεύγουμε κινδύνους. Φυσικά και είναι επικίνδυνη η κατάσταση μερικές φορές, οπότε δεν μπορεί να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει συγκεκριμένης γραμμής ε, και απόλυτης χρηματοδότησης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε στους κινδύνους, να τους αντιμετωπίζουμε. Και χρειάζεται να μας βοηθάτε να διευκολύνουμε τα προγράμματα και όχι αστυνόμευση. γιατί μόνο αν έχουμε ευελιξία μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μερικές φορές, σας είπα, να αρμίξουμε σε κάποια ευκαιρία, άλλες φορές πάλι όχι να κάνουμε πίσω. Τι άλλο, υπάρχει συζήτηση για το τι θα έπρεπε να είναι ακριβώς το καπιστευματικό ταμείο. Θα πρέπει να είναι μια μετάβαση. Να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποια επίγουσα ανάγκη αλλά να μην το βλέπουμε μόνο σαν αυτό και στη συνέχεια να είναι πρόβλημα. Στα προγράμματα που έχουμε βορειοανατολικά, κάτι το οποίο κάναμε είναι φτιάξαμε κάποια κέντρα διατησίας κατά κάποιο τρόπο για να αντιμετωπίσονται προβλήματα βία σε βάρος των γυναικών, σε καταβλισμούς όπου με τον ένα τον άλλο τρόπο υπάρχουν τέτοια προβλήματα βία σε βάρος των γυναικών. Είναι επίγουσα βοήθεια, αλλά αντιμετωπίζοντας αυτή την επίγουσα βοήθεια δημιουργούνται οι κατάλληλες δομές, οργανωτικές, διαχειριστικές, για την παρετέρω ανάπτυξη αυτών των κέντρων. Δηλαδή συγχρόνως φροντίζουμε και μια φιλοδοξία πιο μακροχρόνια για να αντιμετωπιστεί αυτή η βία σε βάρος των γυναικών. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της μεταβατικής ε, παρέμβασης επίσης έχει μεγάλη σημασία για ένα από τα άλλα ζητήματα. Είναι παραδείγματος χάρη η επιτυχής ε, χρήση διάφορων προγραμμάτων. Παραδείγματος χάρη κάποιοι άνθρωποι ε, αναδιατύπωναν τα προγράμματα για να πάρουν νέα χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας δίνει ακριβώς ε, ένα μάθημα για το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα διδάγματα σε νέες ε, συνθήκες. Κάτι το πολύ σημαντικό. Το τέταρτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι η αναγκαιότητα να αντιλαμβανόμαστε το πλαίσιο σε κάποιους ε, τομείς, οπωσδήποτε σε κάποιους από τους που το κράτος, το κεντρικό νιγηριανό κράτος ή το τοπικό κράτος ε, στα βόρειο-ανατολικά απουσιάζει όσον αφορά τις σχέσεις που οικοδομούμε με τις κοινότητες, με άτυπες ή παραδοσιακές δομές. Κάποιοι ίσως το θεωρούν αυτό ως πρόβλημα, ως εμπόδιο. Αλλά εμείς ε, θα λέγαμε το αντίθετο. Είναι μια ευκαιρία για ένα διαφορετικό πρόγραμμα που μας επιτρέπει ακριβώς ε, να κάνουμε αλλαγές μέσω των δομών που υπάρχουν εκεί. Και ηρωνικό είναι το ότι ε, υπάρχει η δυνατότητα σε ανθρώπους περιθωριοποιημένους να αρχίσουν να μιλάνε με το κράτος για αυτά τα οποία χρειάζονται. Οπότε ε, επιτελούμε μια σημαντική λειτουργία με το να μην πηγαίνουμε στον επίσημο κρατικό νομών. Το πέμπτον αφορά τον ε, συντονισμό. Ε, πολλή συζήτηση έχει γίνει. Εμείς θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να εμφανιστεί ο συντονισμός ως διαμαγείας από διαφορετικά προγράμματα. Πρέπει να έχει προγραμματιστεί ευθύ εξ αρχής και ο τρόπος ε, να γίνει αυτό είναι ακριβώς ε, να υπάρχει δυνατότητα αυτή ε, στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα το περιβάλλον αλλά και μπορούν να εργαστούν μέσω αυτών των δομών. Δηλαδή όταν επιβάλλουμε κάτι από πάνω κατά κανόνα είναι μετά κάτι το τυπικό και δεν σημαίνει καθόλου συντονισμό στην πράξη. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το θέμα παρακολούθησης, αξιολόγησης ε, των ε, δίδαγμάτων και αυτό το οποίο αποφεύγουμε, το πώς, ε, το τι ακριβώ είναι η βέλτιστη χρήση των κοντιλίων. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογούμε και να έχουμε κάποια λογικά στοιχεία μέτρησης ε, για το τι κάνουμε μέρα-μέρα, μήνα-το-μήνα, για το πώς χρησιμοποιούμε τα κονδύλια και έτσι με κάποιον ε, τρόπο να βοηθήσουμε και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο. Οπότε, θα έλεγα πως ε, τα καταπιστεύματα αυτά είναι πολύτιμο εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο εργαλείο, αλλά είναι μια αφετηρία. Και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και κατεπίγουσες καταστάσεις, αλλά και μεταβατικές ε, περιόδους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τα πρακτικά αυτά παραδείγματα. Αυτά πρέπει να ακούμε, γιατί αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε τα νέα μας <coughs> προγράμματα και ε, την, ε, τα νέα μας μέσα και ένα θέμα ακριβώ είναι η ευελιξία. Και βεβαίω ακριβώς ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει συνεργασία με τις οργανώσεις επιτόπου και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε περισσότερο. Ξέρω πως είναι η Κομισιόν εδώ Το έχουμε θίξει πολλές φορές ε, και μια που είναι εδώ πέρα και ο υπουργό από τον Ήγηρα. Πριν από 15 μέρες είχα μια κρόαση με την Επιτροπή για τα θέματα της μετανάστευσης στον Ήγηρα και ένας από τους ομιλητές μίλησε ε, μία βουλευτής για τις γυναίκες από την Νιγηρία που είχαν υποστεί την βία του Μπόκο Χαράμ κατέφυγαν στον Νίγηρα και μας είπε ότι επισκέφθηκε τα στρατόπεδα προσφύγων, ήταν άθλια η κατάσταση, ζούσαν ε, σε καθεστώς φόβου. Ε, πραγματικά οφείλουμε να επενέσουμε τη δουλειά που γίνεται και τον Υπουργό γιατί και ο Νίγηρας αντιμετωπίζει προκλήσεις και μετά έχουν και την πρόκληση των ανθρώπων που έρχονται από την Νιγηρία Επίσης είχαμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης, συζητήσαμε τους γάμους ανηλίκων ε, στον ε, Νίγηρα. Βλέπω πως γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και θα ήθελα και οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα να ακούσουν τα όσα είπαν εδώ οι ομιλητές για το τι συμβαίνει. Γιατί ακριβώς πρέπει να αντιληφθούμε το μέγεθος της ε, πρόκλησης αλλά και τη δουλειά που γίνεται επί τόπου και στον Νίγηρα και αλλού. Λοιπόν, κύριε Αρτουή, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ενδιαφέραν πολύ οι μαρτυρίες των εμπειρογνωμόνων, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στα όσα μας είπε ο Υπουργός ε, Μασούντου. Μας είπατε ότι πραγματικά υπάρχει μια εγκληματική οικονομία που οργανώνει τη μετανάστευση κατά κάποιο τρόπο και ότι θα ήθελε να ενισχυθούν οι κρατικές δομές ε, σίγουρα για να προσπαθήσει να περιορίσει αυτή την ε, εγκληματική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, ποια εκτίμηση εσείς κάνετε τις δράσεις της Ευρώπης που αντιναπτύσσεται ακριβώς στην Αφρική. Έχετε προτάσεις, συστάσεις να μας κάνετε τη στιγμή όπου ε, μελετούμε και επεξεργαζόμαστε το επόμενό μας δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ, η Γιάλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να σχολιάσω μόνο σε σχέση με ορισμένα από τις ομιλίες που ακούσαμε και τα, τα όσα ακούσαμε από και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού Έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξαν πολλές συμβάσεις που υπογράφηκαν γιατί πρόκειται για μικροπιστώσεις που δίνονταν στις κοινότητες για να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να μπορέσουν έτσι να αναπτύξουν και να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτές τις καταστάσεις και όπου η Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε τις συμβάσεις, αλλά πολλές φορές δεν έγινε τίποτα. Κάποιες φορές ήταν σημαντικά τα κονδύλια ε, και Στι ακροάσεις μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το θέσαμε πολλές φορές. Ήταν μία από τι επικρίσεις ότι δηλαδή οι μηχανισμοί της ΤΕΠΑ δεν είναι άμεση. Ότι δηλαδή από τη στιγμή που εκκρίνονται αυτά τα προγράμματα για να καταλήξουν τελικά αυτά τα πολύ μικροσκοπικά προγράμματα για την ίδια την τράπεζα, μικροσκοπικά η τράπεζα, αλλά όχι για τις κοινότητες που δέχονταν αυτά τα χρήματα. Ε, περνούσαν ε, πολύ καιρό και κάποιε φορέ δεν φτάνουν ποτέ τα χρήματα. Υπάρχει κάποιο project για να γίνονται λοιπόν και να εφαρμόζονται αυτά τα project. Επίσης, ε, όλα ένα και περισσότερο στις συνεδριάσεις που κάνουμε και αυτό το λέω περισσότερο, εγώ έχω ασχοληθεί περισσότερο με την περιοχή του Μαγκρέμπα, αλλά όχι μόνο οι θύνοντες, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και τα λοιπά οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μια πολιτική σχέση παραπονιούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει να δουλεύει για τις υποδομές, δηλαδή νοσοκομεία, σχολεία και ότι δουλεύουμε περισσότερο για την άλλη αξία, δηλαδή διακυβέρνηση, αξίες και τα λοιπά, που και αυτά είναι καλά, αλλά στα πρακτικά πράγματα υπάρχει κάποια... Ε, και ξέρουμε ότι έχουμε ανταγωνιστές, έχουμε και πολλά προβλήματα γιατί κάποιες υποδομές που κατασκευάζουν ξέρουμε ας πούμε στη Μαυρτανία στην περίπτωση του λιμανιού ξέρουμε ότι είχε φρικτό αντίκτυπο για το περιβάλλον και το είπαν και οι ίδιοι οι άνθρωποι ε, οι Μαυρτανοί Μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση δηλαδή όπου θα μπορούσαμε να συστήσουμε η Επιτροπή γιατί, συγγνώμη που έφυγα για λίγο γιατί είχα και άλλα πράγματα στην Επιτροπή Αναφορών αλλά θα μπορούσαν ίσως και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να μας απαντήσουν. Γιατί έχω ακούμε όλο ένα και αυτά τα, περισσότερο αυτά τα παράπονα, ότι δηλαδή στην ουσία, στην πράξη αυτά που κάνουμε δεν στηρίζουν τις υποδομές, αλλά κάτι άλλο. Δεν, μπορεί, δεν πρέπει δηλαδή να γίνεται ή το ένα ή το άλλο, θα πρέπει και τα δύο να γίνονται, γιατί είναι πολύ σημαντικά για τις χώρες που πρέπει δηλαδή να επιλέξουν ποια project θα στηρίξουν, αλλά τη στιγμή που πρέπει να το επιλέξουν δεν είμαστε εμείς εκεί. Μάλιστα, ο κύριος Βόν θέλει κάτι να ρωτήσει. Θα σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Και μετά από τα όσα μας είπε η Ίνες, Να υπάρχει, είπαμε, περισσότερη ευελιξία, ναι. Αλλά θα υπάρχουν και συνάδελφοι που θα αρχίσουν να βγάζουν ε, καντήλες όταν θα ακούσουν αυτά για περισσότερη ε, ευελιξία. για την χρηματοδότηση των project, ε, την ε, υλοποίησή τους. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει προσθέμενη αξία χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορείτε αυτό να το δείξετε στην καθημερινή σας δουλειά. Γιατί η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ε, ενδιαφέρεται περισσότερο για την λογοδοσία. Για... Είναι δύσκολο να το επιτύχουμε. Είναι αυτού του είδους ερωτήσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο προπολογισμού. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάθε κόσμο εδώ στις Βρυξέλλες και να αντιληφθεί το τι γίνεται εκεί επί τόπου. Θα ακούσουμε πρώτα τον Υπουργό, γιατί του έγινε μία ερώτηση τον κύριο Αρτουή για το πώς βλέπει την επιτυχία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κύριε Υπουργέ, ε, την ερώτηση και οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε έτσι, συνοψίζοντας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν μίλησα για την ε, εγκληματική οικονομία που αντικατέστησε την επίσημη εξαιτίας ε, της εύθραυστης κατάστασης που υπάρχει κυρίως στο Βορρά. Προσπάθησα να το εξηγήσω πριν. Και η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια χειροτέρεψε πολύ στη Λιβύη. Εξού και το πρόγραμμα με το Δούνου του τότε, τη δεκαετία του 90 δηλαδή, οδήγησε στο να αποσυρθεί η χώρα από επενδύσει στην εκπαίδευση, την υγεία, ακόμα και την ασφάλεια. Και γι' αυτό, έχοντας αποσυρθεί το κράτος, έγιναν ακόμα πιο ασταθείς οι περιοχές της περιφέρειας. Εξού και η οικονομία, η αγροτική, ο τουρισμός που πηγαίνανε καλά πριν, ήταν καλά γιατί υπήρχε ασφάλεια. Το Παρίντακαρ περνούσε από εκεί. Υπήρχαν τσάρτερς που ερχόντουσαν από τη Μασαλία το Παρίσι υπήρχε μια ανθούσα τουριστική οικονομία η οποία ξαφνικά εξαφανίστηκε. Όσο περισσότερο δημόσιες υπηρεσίες εξέλιπαν και οι επενδύσεις οι δεν υπήρχαν, μετά το λαθρεμπόριο σιγαρέτων, ναρκωτικών Τώρα, με την κατάρρευση του κράτους στη Λιβύη, για όποιον λόγο και αν έγινε αυτό, περάσαμε στη λαθροδιακίνηση. Δημιουργήθηκαν δίκτυα δηλαδή που φτιάξανε μια οικονομία η οποία λειτουργούσε. Πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που έγιναν ήταν για την ασφάλεια. Υπήρξαν προγράμματα επίγουσας βοήθειας με το καταπεστηματικό ταμείο. Τα 53 εκατομμύρια, εντάξει, πολύ λίγα χρησιμοποιήθηκαν. Κάποια προγράμματα άρχισαν. Κάποια ελοπίθηκαν γρήγορα. Έγινε αυτό. Αλλά ακόμα και για Άλλε επίγουσες ε, περιπτώσεις αυτά τα 153 εκατομμύρια δεν έχουν καν χρησιμοποιηθεί γιατί οι διαδικασίες είναι βαριές ενώ η επίγουσα βοήθεια πρέπει αμέσως να δοθεί ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι αναμένοντας τις πιο μακροχρόνιες βοήθειες. Όλα αυτά τα ανέλαβαν οι υπηρεσίες εκτέλεσης εκτός κράτους. Γι' αυτό λέω ότι το κράτος πρέπει να αποκτήσει και πάλι τις αρμοδιότητές του. Αυτό είναι που ζητάω. Και αυτό είναι που θα βοηθήσει στη διάρκεια και θα γίνουν και επενδύσεις ε, στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει ότι επιστρέφουν οι δημόσιες υπηρεσίες και ότι θα μπορέσουν έτσι να υπάρξουν προγράμματα με ε, τις κρατικές αρχές και τους διάφορες, ε, τους διάφορες συλλόγους και οργανώσεις. Σε συνεργασία χρειάζεται διάρθρωση με την ανάπτυξη και με τον κύριο φορέα. Πριν έρθει το κράτος να συνδράμει, συγγνώμη, ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει, πρώτα το κράτος. Αυτό είναι που θέλω να πω. Πρέπει να αποκατήσουμε σταθεί το κράτος, να νομιμοποιηθεί και πάλι, γιατί η απόσυση του κράτους από όλα αυτά είναι που στις εγκληματικέ ε, δραστηριότητες και δεν ξέρω αν ε, δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση ο κύριος Σαρτουή. Όταν μιλάμε για εγκληματική οικονομία, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία αυτή χρηματοδοτείται από κάπου από πού προέρχεται η χρηματοδότηση αυτών που συμμετέχουν στην εγκληματική οικονομία, δηλαδή οι μετανάστες, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς πληρώνουν τους ε, εγκληματίες αυτούς. Μα είναι λαθροδιακινητές που έχουν οχήματα. Και ποιος τους πληρώνει, ρωτά ο κύριος ε, Αρτουή. Μα <clears throat> είναι οι ε, λαθρέμποροι ναρκωτικών. Αυτοί είναι που έχουν χρήματα και που ελέγχουν την οικονομία σε όλη αυτή την περιοχή που ξεκινάει από, την, ε, από τον Νότο, περνάει από το Σαχέλ και φτάνει στην Ευρώπη. Η εγκληματικότητα που έχει να κάνει με τους μετανάστες είναι μια δευτερεύουσα, έτσι, απόρρια. Γι' αυτό εμείς στη διάσκεψη στη Λαβαλέτα προτείναμε ένα πρόγραμμα που θεωρήθηκε πολύ φιλόδοξο. Λίγο κάτω από ένα δις φτάσαμε στα 300 περίπου, 314 εκατομμύρια τελικά. Μένουν 90 ακόμα. Πώς να κινητοποιηθούν αυτά. Έτσι καλλιώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα ολόκληρο δίκτυο και να καλύψουν όλους αυτούς που ζουν από τα παράνομα δίκτυα. Ναι, αλλά οι μετανάστες, ρωτά ο κύριος Σαρτουή, είναι οι ίδιοι που πληρώνουν, έτσι δεν είναι οι οικογένειές τους. Ναι, ναι, οι μετανάστες έρχονται με πολλά χρήματα και πληρώνουν στα καντέ, στη Λιβύη και αλλού. Είναι και αυτοί οι μετανάστες που βρίσκουν αυτά τα χρήματα για να πληρώνουν τους εγκληματίες. Στη χώρα προέλευσης, λέει ο κύριος Μασούντου, γιατί βοηθούν οι οικογένειες στις χώρες προέλευσης για να πληρωθεί η μεταφορά αυτή των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρώπη και μετά δημιουργούνται διάφορα δίκτυα ή αν έχουν δουλειά στη μαύρη κτλ. Επιστρέφουν τα χρήματα στις χώρες τους αν ήταν δάνειο ας πούμε. Οι λαθροδιακινητές όμως συμμετέχουν στην, στον Ήγερα, στη Λιβύη και αλλού συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οικονομία, είναι γνωστό. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που είναι απόρρια του λαθρεμπορίου στην περιοχή λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ναι, αλλά οι μετανάστες δεν έχουν λεφτά πάνω τους, λέει ο κύριος Σαρτουή. Υπάρχουν παράλληλα τραπεζικά, ας πούμε, συστήματα. Όχι, λέει ο κύριος Μασούντ, έχουν ρευστό απάνω τους. Δεν ξέρω, όχι, έχουν ρευστό. Μα έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις, τα βλέπουμε αυτά. Ρευστό κυκλοφορεί τώρα, και αυτό είναι πρόβλημα σε σχέση με την εγκληματική οικονομία. Θα έπρεπε να περνάνε μέσα από την τράπεζα. Στον Ήγερα, για παράδειγμα, μόνο 6% για να έρθω στην ερώτηση για τις μικροπιστώσεις της κυρίας. Μα πρέπει να υπάρχει μικροχρηματοδότηση για να, υπάρχει, να υπάρχουν μικροπιστώσεις. Και το λέω αυτό για να καταπολεμήσουμε ακριβώς όλη αυτή τη ροή χρήματος παράνομου στο τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την κυκλοφορία του ρευστού χρήματος και να αυξηθεί το ποσοστό του χρήματος που περνάει μέσα από τις τράπεζες. Το ρευστό κυκλοφορεί. Γι' αυτό θα οργανώσουμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά την ερώτησή σας. Ξέρω ότι έχει συμφωνίε ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με διάφορες ε, τράπεζες για μικροπιστώσει, Δεν έχει λειτουργήσει όμως. Συζήτησα και εγώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να συμμετέχει σε μία στρατηγική μας. Θα έχουμε μία διάσκεψη ώστε όσοι θέλουν να στηρίξουν τη στρατηγική μα για μικροπιστώσει, να το κάνουν είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά είναι και ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπιστεί η εγκληματική οικονομία. Η ανακύκλωση αυτή του παράνομου χρήματος. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Πρόεδρος. Μα ναι, διευκρινίσατε, απαντήσατε στις ερωτήσεις, οπότε αυτό θέλαμε και από εσά έτσι κι αλλιώς. Οπότε μην ζητάτε συγγνώμη. Λοιπόν, Μπομπ. Θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην ερώτηση αυτή που έγινε για το πού βρίσκουν τα χρήματα οι μετανάστες. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε, στα σύνορα του Νίγηρα υπάρχει τεράστια κρίση εξαιτία του Μπόκο Χαράμ. Και οι μετανάστες δεν είναι από την βόρειο-ανατολική, από το βορειοανατολικό Νίγηρα. Είναι άνθρωποι από άλλες χώρες ε, νότια του Νίγηρα που βλέπουν τη μετανάστευση σαν οικονομική ευκαιρία και τους χρηματοδοτούν οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους, γιατί αν έχουν ένα συγγενή οικογένεια στην Ιταλία, τέλος πάντων κάπου στη Δυτική Ευρώπη, πρώτα απ' όλα θα τους στέλνει εμβάσματα και δεύτερον αυξάνει την ευκαιρία και για αυτούς. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία μετανάστευση για αυτού του είδους των μεταναστών που δεν είναι βέβαια όλοι έτσι. Το θέμα της ευελιξίας. Έχουμε τώρα μια κατάσταση όπου μπορούμε να ξοδεύουμε παραδείγματο χάρη στην τεχνική αρρωγή, αλλά δεν μας επιτρέπεται να ξοδέψουμε σε υποδομές. Έρχονται λοιπόν οι Νιγηριανοί εταίροι και θέλουμε να έχουμε, όπως μας είπατε, ένα ε, δικαστήριο για οικογενειακές υποθέσεις και εμείς λέμε ναι θα κάνουμε τεχνική αρρωχή και μας λένε «Μα δεν έχει οροφή το κτίριο». Και τους λέμε «Α, υποδομές ε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε». Αλλά δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δώσουμε και την τεχνική αρρωγή μετά. Δηλαδή αυτά είναι έτσι μια ευελιξία μικρής ε, κλίμακας ε, που θα μας έδινε την δυνατότητα τελικά να δώσουμε και την τεχνική αρρωγή. Για το θέμα των μικροπιστώσεων. Ορίστε. Ένα από τα θέματα που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι συχνά οι συμφωνίες υπογράφονται με λάθος ανθρώπους. Δηλαδή, δεν έχει πάει η διαπραγμάτευση σε βάθος έτσι ώστε τα άτομα τα οποία θα λαμβάνουν τη μικροχρηματοδότηση να είναι στην συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει κανεί με τον Υπουργό Οικονομικών, με τα υψηλά κλιμάκια τη Νιγηριανή κυβέρνηση που θα εγκρίνουν πολλά πράγματα. Αλλά το εάν αυτό τελικά θα φτάσει στου ανθρώπου στην ε, κοινωνία είναι κάτι το τελείω διαφορετικό. Τέλο, Το θέμα που ετέθη ή για το εάν ε, μπορούμε να δώσουμε κάποια ασφάλεια όσον αφορά την χρηματοδοτική ευελιξία και το εάν θα χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια. Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν ε, τα προγράμματα εκεί πέρα έχουμε κάποιες ε, σοβαρές οργανωτικές δομές. Όταν αναλαμβάνουμε έργα με τους εταίρους μας στην Ιγυρία δεν εκταμιεύουμε τεράστια ποσά την πρώτη εβδομάδα και αναμένουμε να γίνει το έργο, γίνεται με δόσεις, με αποτελέσματα, να γίνεται μεγάλος έλεγχος. Κάνουμε λάθη, ναι, κάνουμε λάθη βεβαίως. Νομίζω πάνω από 90% τα κάνουμε σωστά και αν δεν αναλάβουμε αυτό το ρίσκο θα καθόμαστε πάνω στα λεφτά τα οποία δεν θα επιτύχουν την ανάπτυξη την οποία θέλουμε. Και το τελευταίο ζήτημα το οποίο ήθελα να αναφέρω αφορά αυτό το θέμα του κράτους. Σαφώς είναι ένα θέμα πλαισίου. Σε κάποια σημεία το κράτος και όπως στην βόρειο-ανατολική Νιγηρία έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση το κράτος και δεν έχει νόημα να συνεργαζόμαστε και με το κράτος. Εκεί όπου έχει μια στιβαρή παρουσία και νομιμοποίηση είναι βεβαίως, κάντε το. Αλλά το ερώτημα είναι να μην έχουμε ε, ένα καλούπι και να λέμε πρέπει να περάσετε από το Υπουργείο. Να αναγνωρίζουμε το πλαίσιο και τις διαφορετικές συνθήκες. Μάλιστα. Ε, είπατε, δώσατε το παράδειγμα του δικαστηρίου. Ότι δεν μπορείτε να κάνετε έργα υποδομής. Ε, και δικομισιών, οι ειδικοί έφυγαν ε, ίσως μπορούμε να ζητήσουμε την Κομισιό να μας απαντήσει μια άλλη στιγμή. Ποιος αποφασίζει αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή μπορείτε να χρηματοδοτήσετε αυτό, ε, τεχνική αρρωγή ας πούμε, αλλά όχι υποδομές. Ποιος θα αποφασίσει. Είναι οι Βρυξέλλες. Είναι η αντιπροσωπεία γιατί τώρα ξεκινάει η συζήτησή μας για τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τη νέα γενιά ε, ταμείων και αν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα πρέπει να τα λύσουμε. Τώρα είναι η ευκαιρία αν υπάρχουν ε, προβλήματα, αν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν για την χρηματοδοτική στήριξη. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε κάποιες χώρες και υπάρχει επιφυλακτικότητα από τους συναδέλφους του του προπολογισμού για την στήριξη του προπολογισμού, αλλά σε άλλες χώρες λειτουργεί. Όπως είπατε, ναι, ο καθένας και κατά περίπτωση δεν είναι ένα ενιαίο καλούπι. Δεν ξέρω, η Κομισιόν τώρα που ίσως μπορεί να έρθει μια άλλη φορά και να μας πει τι γίνεται με το καταπίστευμα, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί, γιατί σε έναν ιδεώδη κόσμο θα υπήρχε μια διάρθρωση μεταξύ καταπιστευμάτων, ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα πηγαίνουν σε διαφορετικά, κινούνται σε ε, διαφορετικούς άξονες. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε γρήγορα. Να έχουμε κάποια λεπτά ακόμα. Κυρία Μπεχάρη, θα ήθελα να αντιδράσω γιατί ακούστηκαν ε, πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και από τον Υπουργό Οικονομικών αλλά πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά δεν επαρκούν πως ακριβώς αναφέρθηκε και ο κύριος υπουργό και νομίζω πως ε, δεν σπάνε τελικά οι δίωδοι των ε, λαθροδιακινητών απλά γίνονται πιο ακριβοί οπότε η πραγματική αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να πάει στις ε, πραγματικές ανάγκες καταπολέμηση της φτώχειας κτλ και όταν μιλάμε για τη μετανάστευση πρέπει να δεχτούμε το ότι η μετανάστευση είναι τμήμα της ανθρώπινης βύσης, να κάνουν προγράμματα βίζας, ε, όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών αλλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε εργασία, έχουμε χώρο ε, και επίσης οι αιτούντες άσυλο να μην πεθαίνουν στην θάλασσα, να μην χρειάζεται να πληρώνουν κανέναν, ε, να είναι θύματα διακινητών ή σκλαβιά στη Λιβύη αλλά να φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανθρωπιστικές βίζες οι οποίες ε, θέλει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Επίσης ε, έχω αναφέρει κάποια ζητήματα τη επαναγκατάσταση και εναλλακτικών διόδων που είναι απαραίτητα για πρόσφυγε και μετανάστες και σα ευχαριστώ που μου δώσετε τον λόγο. gonna... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Βόν για να ολοκληρώσει την συνεδρίαση. να πω και εγώ ευχαριστώ στο επιτελείο μας και στη γραμματεία των Επιτροπών που διοργάνωσαν τη σημερινή ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τη συμβολή του και φυσικά όλους μας τους εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ καλό μείναμε εδώ και εργαστήκαμε γιατί ε, πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε από πρώτο χέρι αυτού του είδους τις λεπτομέρειες, γιατί θα αρχίσουμε να τώρα να συζητάμε και το επόμενο ε, πλαίσιο αλλά θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τις λεπτομέρειες των επομένων προγραμμάτων. Οπότε όσο περισσότερες συζητήσεις κάνουμε, τόσο περισσότερο θα μάθουμε και ως βουλευτές για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στον επόμενό μας προϋπολογισμό, να δούμε τι είναι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν που ήρθατε και εμείς σίγουρα θα τα λάβουμε υπόψη τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ. Τέλος της συνεδρίασης. Και ευχαριστούμε και τους ομιλητές μας βέβαια.